Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ για τους ομιλητές που βρίσκονται εδώ και ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Γίνονται πολλά έργα στις υδροδρομικές γραμμές ε, γύρω από τις Βρυξέλλες. Προτείνω να ξεκινήσουμε ευθύ αμέσω με το σημείο 1. Να υπενθυμίσω πρώτα απ' όλα τους ε, γλωσσικούς κανόνες ε, για την υποεπιτροπή μας θα σας ε, παραθέσω τις γλώσσες που δεν μεταφράζουμε σήμερα το πρωί. Βουλγάρικα, τσέχικα, κροατικά, δανέζικα, ολλανδικά, φιλανδικά, ιρλανδικά, λετωνικά, μαλτέζικα, πορτογαλικά, σλοβάκικα, σλοβένικα και σουηδικά. Στις υπόλοιπες γλώσσες υπάρχει διερμηνία. Δεν έχουμε ιδιαίτερε παρατηρήσει για την ημερήσια διάταξη, μάλλον, οπότε μπορούμε να εγκρίνουμε τη σημερινή ημερήσια διάταξη. Ανακοινώσεις της Προεδρίας, να σας υπενθυμίσω, 21 Νοεμβρίου, μεταξύ 11.30 και 1 θα έχουμε μια έκτακτη συνεδρίαση αυτής της Επιτροπής ε, με την παρουσία του κυρίου Ζαν Πιέρ Λακρόα, αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα των ΟΕΕ για τις ε, ειρηνευτικές επιχειρήσεις. Έκτακτη λοιπόν συνεδρίαση της ΣΕΝΤΕ από κοινού με τις ΑΦΕΤ και ΝΤΡΟΑ. 5η 21 Νοεμβρίου από τις 11 και μισή μέχρι τη μία. Άλλες ανακοινώσεις όσον αφορά τις, ε, τις συνεδρίες των συντονιστών και τις σχετικές αποφάσεις της 25 Σεπτεμβρίου του 2019 σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό τα συμπεράσματα έχουν ανέβει στην ιστοσελίδα της ΣΕΝΤΕ όπως και τα υπόλοιπα έγγραφα της συνεδρίας αυτής και επισυνάπτονται στα πρακτικά της συνεδρίασης 25ης και 26ης Σεπτεμβρίου. Όσον αφορά τα πρακτικά συνεδριάσεων, ε, τη συνεδρίαση της 9 η ε, Σεπτεμβρίου, της 25ης, της 26ης Σεπτεμβρίου και της 8ης Οκτωβρίου έχουν διανεμηθεί. Αν δεν υπάρχουν ιδιαίτερα σχόλια, να τα εγκρίνουμε. Σας ευχαριστώ. Πάμε τώρα στην ακρόαση για την ασφάλεια και την άμυνα στο διάστημα. Θα γίνει μια ανταλλαγή απόψεων με τους προσκεκλημένους μας, ε, τους οποίους ευχαριστώ ξανά, Ολιβιέ Ζαγιέκα, Διευθυντής του Ιδρύματος Μελετών και Στρατηγικής και Άμυνας, ε, παιδαγωγικός υπεύθυνος στο Μάστερ 2 για την ασφάλεια και την άμυνα διεθνώς ε, στην νομική του Πανεπιστημίου Ζάμουλα Λιον 3, Πασκάλ ε, επικεφαλής επιχειρήσεων της GSA, η κυρία Καρίν Κλέης, ε, ειδική επεσταλμένη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διάστημα και η κυρία Σιμονέτη Ντίπιπο, διευθύντρια UNOS ε, των Ηνωμένων Εθνών. Αγαπητοί συνάδελφοι, εκ μέρους της Υποεπιτροπής μας θέλω να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους που ήρθαν εδώ να μας μιλήσουν Σήμερα θα ήθελα να ξεκινήσουμε αυτό που ονομάζω εγώ έναν κύκλο για το διάστημα. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει σημαντικά στον τομέα του διαστήματος. Οι ιδιωτικοί φορείς όλο και περισσότεροι ε, έχουν πλέον ε, διαστημική παρουσία και νέοι επίσης κρατικοί φορείς ε, έχουν μια νέα παρουσία. Ο τομέας εξελίσσεται με τεράστια ταχύτητα και μεγάλο εύρος. Είναι εντυπωσιακό οι οικονομίες, οι κοινωνίες μας, οι υποδομές μας, δημόσιες και οι δημόσιες υπηρεσίες μας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το διάστημα. Το ίδιο και τα πολιτικά μας συστήματα και οι στρατιωτικές μας δραστηριότητες. Όλα αυτά εξαρτώνται από τις δορυφορικές επικοινωνίες. Έτσι λοιπόν το διάστημα είναι στρατηγικός κόμβος ύψης της σημασίας για τις αναπτυγμένες κοινωνίες μας. Όλες εξαρτώνται από αυτό και ευάλωτες ε, σε περίπτωση προβλήματος. Οπότε το να λαμβάνουμε υπόψη το διάστημα στα θέματα άμυνας και ασφάλειας είναι κάτι αναγκαίο. Οι ΙΠΑ έχουν ξεκινήσει ε, ένα επιτέλειο για το διάστημα. Εδώ το ξεκινάμε εμείς στα κράτη-μέλη επίση και εδώ στην Επιτροπή μας θέλουμε να ενημερώνουμε για τις διεθνείς συνθήκε στον τομέα του διαστήματος και τη θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη δεν ε, μπαίνει σε έναν πόλεμο των άστρων αυτή τη στιγμή, ούτε Όμω πρέπει να καθυστερεί όσον αφορά την επιτήρηση του διαστήματο και την προστασία των δορυφορικών μα συστημάτων. Η θέση τη Ευρώπη στον νέο, διαστημικό αγώνα δεν είναι βέβαιη. Εάν σημειώσουμε καθυστέρηση θα είναι δύσκολο να την καλύψουμε. Ευτυχώ η, πρόεδρο τη Επιτροπή, ε, εξέφρασε την πρόθεση να δημιουργήσει μια γενική διεύθυνση που θα συγκεντρώνει τι βιομηχανίε άμυνα και διαστήματο και στο επόμενο πολιτισμό δημοσιονομικό πλαίσιο προβλέπουμε την ε, ανάλογη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής ε, Διαστημικής Πολιτικής. Όλο και περισσότερες απειλές εμφανίζονται στο διάστημα, τα διαστημικά απόβλητα, θέμα που μας αποσχολεί εδώ και γερό και που ε, γίνεται όλο και σημαντικότερο οι απειλές του κυβερνοχώρου αλλά και οι κακόβουλες συμπεριφορές εχθρικών στρατιωτικών δορυφόρων δίπλα στους δικούς μας δορυφόρων Μία λοιπόν ευρωπαϊκή πολιτική διαστημικής άμυνας φαίνεται να είναι κάτι επιβεβλημένο. Βάσει όλων αυτών θα ήθελα να ξεκινήσουμε δίνοντας πρώτα απ' όλα το λόγο στον κύριο Ολιβιέ Ζάιεκ. Ε, είστε διευθυντής του Ιδρύματος Μελετών Στρατηγικής και Άμυνας. Είστε επίσης ε, εκπαιδευτικός υπευθυνός σε ένα μάστερ στο Πανεπιστήμιο Ζωμουλά στη Λιόν Επιφορτισμένο με τα μαθήματα γεωπολιτική στη Σχολή Πολέμου στο Παρίσι από το 2015 και ο ελέκτρο στο Ίδρυμα Υψηλών Σπουδών Εθνικής Άμυνας και στο Κέντρο ε, Ανώτατων Στρατιωτικών Σπουδών. Θα μας ε, παρουσιάσετε μια εικόνα των γεωπολιτικών προκλήσεων που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μπροστά σε αυτό που θα ονομάζαμε στρατιωτικοποίηση του διαστήματος και θα μας μιλήσετε για τις ε, επενδύσεις και τα ε, πρακτικά θέματα για τις χώρες εταίρους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, να ευχαριστήσω την Υποεπιτροπή Θεμάτων Άμυνας για την πρόσκληση αυτή. Είναι τιμή για μένα να σας απευθύνω το λόγο για ένα σημαντικό θέμα για την Ευρώπη. Εξαιρετικά ευρύ θέμα και αναγκαστικά σε 10 λεπτά θα πρέπει πολύ συνοπτικά να τοποθετηθώ. Ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων και ζητώ συγγνώμη και από τους διερμηνείς, αν είμαι ταχύς, λέει ο μιλητής. Λοιπόν, έχουμε έναν ανταγωνισμό εξοπλισμών ε, άνω της ατμόσφαιρας και αυτό δεν ε, περιορίζεται μόνο στις ε, τεχνολογικά προηγμένες χώρες και πρόκειται για μια τάση πολύ έντονη, διότι αυτό που παρατηρούμε δεν περιορίζεται στην ε, πολιτική δραστηριότητα. Έχουμε μια διτή στόχευση των επενδύσεων στο διάστημα και όλα αυτά ενέχουν μια διάσταση στρατιωτική, είτε άμεση είτε έμεση και η στόχευση αυτή πρέπει να, μάλλον αυτή υφίσταται είτε αναγνωρίζεται είτε δεν αναγνωρίζεται από τα κράτη επισήμως. Επομένως σε μια πρώτη ανάγνωση μπορούμε να μιλήσουμε για εκδημοκρατισμό του διαστήματος. Αλλά όχι μόνο σε επίπεδο τεχνολογικό ή προόδου τεχνολογικής για την καθημερινή μας ζωή, αλλά προόδου στρατιωτικής και αμυντικής. Είτε μάλιστα επιθετικά, είτε αμυντικά σε επίπεδο εξοπλισμού. Επομένως, τα πιο σημαντικά κράτη του 21ου αιώνα ε, θέλουν να θεσπίσουν αυτή την τέταρτη, το τέταρτο πεδίο στρατηγικών εξοπλισμών εκτός από τις χερσαίες θαλάσσιες και αέριες ε, δυνάμεις και ακριβώς θέτουν αυτή την τέταρτη δύναμη, τη διαστημική, ε, σε ισότιμο επίπεδο με τις υπόλοιπες. Επομένως έχουμε μια εντατικοποίηση γενικευμένη των φιλοδοξιών των διαστημικών. Μπορεί λοιπόν κανείς να θεωρήσει ότι το πεδίο αυτό, όπως λένε κάποιοι αναλυτές, ε, προχωρεί προς κάποια εξομοίηση, εξίσωση, όπου ίσως κάποιες χώρες πιο καθυστερημένες θα μπορούσαν να προλάβουν τους πιο προηγμένους. Θεωρώ ότι επ' αυτού ε, θα πρέπει να είμαστε κάπως επιφυλακτικοί. Για τα νέα χαρακτηριστικά αυτού του πεδίου του υπέρ της ατμόσφαιρας ήθελα να σημειώσω δύο στοιχεία. Πρώτον, ε, το διάστημα Ε, γνωρίζει αυτή τη στιγμή μία ε, με, μία ορμή και δεν μπορεί να περιοριστεί σε αυτό που ε, ονομάζουμε σήμερα new space, νέο διάστημα, νέο χώρο. Υπάρχει λοιπόν μία ανατροπή και βλέπουμε πάρα πολλούς νέους δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς φορείς να είναι ενεργείς σε αυτόν τον χώρο, σε αυτό το πεδίο, το οποίο όμως δεν σημαίνει ότι ανατρέπονται οι παραδοσιακές ε, στρατιωτικές και στρατηγικές ιεραρχίες. Η πρόεδρος το υπογράμμισε ήδη προηγουμένως. Αυτά, ε, η τάση αυτή ενισχύεται γεωμετρικά εδώ και μία δεκαετία αλλά επαναλαμβάνω πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και επιφυλακτικοί, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στους αμυντικούς εξοπλισμούς. Η πολυμέρεια εδώ ε, δεν σημαίνει αναγκαστικά και ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού για τους διάφορους φορείς. Υπάρχει λοιπόν αυτή η τάση, μια διπλή τάση και συνέχειας και ρήξης. Καταρχά υπάρχουν οι νέοι παίκτε, όπω θα μπορούσε να του αποκαλέσει κανεί. Το στρατιωτικό επίπεδο φαίνεται ιδιαίτερα ενεργητικό για την περιοχή της Ασίας. Είτε η Ινδία, είτε η Κίνα, είτε η Ιαπωνία, είτε οι υπόλοιπες ισχυρές χώρες, η Νότιος Κορέα, η Αυστραλία, το Πακιστάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Σιγκαπούρη, το Ιράν, και άλλες χώρες πέραν ε, των χωρών που έχουν ήδη μια ικανότητα πυραυλική όπως η Βόρειος Κορέα, το Ισραήλ και το Ιράν. Το Τελαβίβ ήδη έχει ένα σεληνιακό πρόγραμμα και συνεργασία με τους Αμερικανούς και τους Ινδούς δεν έχει καμία διάθεση να παραχωρήσει ε, οποιαδήποτε πλεονέκτημα, οποιαδήποτε δυνατότητα στο Ιράν. Το 2003 ε, το Ιράν δημιουργήσε διαστημική υπηρεσία με ένα ανώτατο συμβούλιο για το διάστημα υπό το Υπουργείο Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Τον Ιανουάριο του 2019 οι ερευνητές του Ιράν δηλώνουν ότι το Ιράν προχωρεί προς την κατάκτηση του τελευταίου αυτού μετόπου, του διαστήματος δηλαδή. Και είχαμε και τον δορυφόρο ΟΜΙΔ ε, που ετέθησε τροχιά το 2009. Για τη Βόρεια Κορέα ε, παρακολουθήσαμε όλη τη διαπραγματεύση μεταξύ του Κιμ Ζονγκούν και του πρόεδρου Τραμπ και μιλούμε για την βαλιστική δυνατότητα, αλλά υπάρχει και μια διαστημική ε, ε, διάσταση. Μεταξύ του 2006 και του 2012 είχαμε ένα πρώτο ρηφόρο του, της Βορείου Κορέας ε, και μάλιστα με αυτόνομη θέση σε τροχιά του δορυφόρου αυτόρου με, χρησιμοποιώντας τον βαλιστικό πύραυλο Taipong 2 θα μπορούσε η Βόρειος Κορέα να βελτιώσει πολύ τις τεχνολογικέ της δυνατότητες τα επόμενα χρόνια. Οι υπόλοιπε ασιατικέ χώρες δεν έχουν άμεση επιθυμία ε, πυραυλική ή δορυφόρων, αλλά η Αυστραλία η οποία δεν έχει διαστημική υπηρεσία, μάλλον δεν είχε μέχρι πέρυσι, ε, ε, δηλώνει πλέον ότι μέχρι το 2030 θα διπλασιάσει το προσωπικό της σε αυτό το τομέα. Η Νότιος Κορέα μόνο το 2006 εκκίνησε στην, ε, στο πεδίο αυτό, διεκδικώντας μια αυτόνομη στρατηγική ικανότητα και έχουμε και μια τελείως διακριτή χώρα. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μελετήσει πολύ προσεκτικά τι κάνει η Σιγκαπούρη, το τοπικό τεχνολογικό πεδίο ε, ε, προοδεύει ε, συνεχώς αναπτύσσεται συνέχεια από το 2012 με μικροδορυφόρους που τίθενται σε τροχιά εκμεταλλευόμενοι την ευνοϊκή του θέση κοντά στον Ισημερινό. Υπάρχουν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που έχουν θέσει μια πρώτη εκτόξευση δορυφόρου σε τροχιά γύρω από τον Άρη, μια αποστολή για, το, για τα επόμενα χρόνια. Υπάρχει όμως μια πολύ έντονη κινητικότητα και στην στρατιωτική διάσταση, στην αμυντική διάσταση και επιθετικός και αμυντικός να εξελίσσεται συνέχεια. Στη Νότιο Αμερική θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και τη Βραζιλία αλλά θα ήθελα να προχωρήσω λίγο περισσότερο. Τώρα, αυτές οι νέες δυνάμεις ε, χρησιμοποιούν τους δικούς τους δορυφόρους και η ανάπτυξη των αμυντικών τους προγραμμάτων είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη παρότι έχουμε πολλές χώρες συνήθως εξαρτώνται από την πυραυλική ή εκτοξευτική ικανότητα άλλων. Ε, συνήθως οι Αμερικανοί, οι Ρώσοι και οι Ινδοί σημειώνουν τις πιο σημαντικές πρόοδους αυτό το new space που λέμε μπορεί να φαίνεται ως εναλλακτικό πεδίο για αυτούς τους νέους παίκτες, αυτές τις νέες χώρες. Ίσως θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ένα new space καινοτομία, ανταγωνισμού, ε, πεδίου αντιπαράθεσης μεταξύ κρατών. Όμως παρότι έχουμε νέους ιδιωτικούς φορείς ιδιαίτερα από τις ΗΠΑ, διατηρούν αμυντική σχέση πολύ έντονη με την Ουάσιγκτον και με τις... Ε, ε, με την, αν θέλετε, με το πεδίο πελατών της. Έχουμε πολλούς κρατικούς φορείς όμως στην Ασία, στην Αφρική, στην Αμερική, νέες διαστημικές υπηρεσίες και φορείς. Όλα αυτά θα προχωρήσουν με τον εκδημοκρατισμό που σας έλεγα αυτού του χώρου του διαστήματος που προς το παρόν είναι υπό απόλυτη κυριαρχία της Δύσεως. Όλα αυτά θα εξαρτηθούν και από τις ευκαιρίες για τον ιδιωτικό τομέα, αλλά όλοι αυτοί οι φορείς προσπαθούν να ενισχύσουν την στρατηγική τους αυτονομία. Οι πραγματικέ ρήξεις και τα ποιοτικά άλματα ως προς την διαστημική ανάπτυξη, που κυρίως ενδιαφέρουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, προφανώς εξαρτώνται από τους κυρίαρχους παίκτες στο πεδίο του διαστήματος. Το νέο αυτό πεδίο του διεθνούς διαστήματος είναι υπό τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία, την Ιαπωνία, την Ινδία και την Ευρωπαϊκή Ένωση ως πιο ισχυρούς παίκτες και μιλούμε για τον ανταγωνισμό και τους σχετισμούς δυνάμεων μεταξύ αυτών των πιο ισχυρών παικτών που ελέγχει αν θέλετε τα, τις κινήσεις ε, των ε, κομματιών σε αυτό το τεράστιο παιχνίδι σκάκι στο διάστημα. Ε, στην Ασία, υπό την έννοια των παραδοσιακών δυνάμεων, έχουμε η Ινδία και η Ιαπωνία, που είναι οι χώρες που ηγούνται σε αυτήν τη διαστημική προσπάθεια οι δευτερεύουσε δυνάμει αν μπορούμε να τις πούμε έτσι, καλούνται να ευθυγραμμιστούν υπό τις περιφερειακές ισχυρές δυνάμεις που υποστηρίζει το Τόκιο και το Πεκίνο επίσης. Η Asia Pacific ε, Space Cooperation υπό την ε, Ινδία και η αντίστοιχη συμμαχία υπό την ε, Ιαπωνία. Η Ινδία αρνείται αυτόν τον διπολισμό μεταξύ Πεκίνου και Τόκιο και προσπαθεί να εισέλθει ως ε, κυρίαρχο στρατηγικός παίκτης. Έχουμε, έχουν σημειωθεί ε, έντονες προοδοί με δύο δορυφόρους ε, παρατήρησης ε, που έχουν εκτοξευθεί από την Ινδία και με δοκιμές αντιδορυφορικών επιχειρήσεων και όλα αυτά δίνουν ένα ισχυρό σήμα της έντονης αυτής ε, προόδου της στρατιωτικής, ε, διαστημικής στρατιωτικής της Ινδίας. Επίσης ε, φαίνεται να έχει μια επιθετική νέα τάση η Ρωσία. Χρησιμοποιεί συστήματα αντιμετώπισης στο GPS, το έχει κάνει και στον Donbass και συστήματα laser κατά των δορυφόρων. Πώς λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει υπόψη τη σήμερα όλη αυτή την κινητικότητα, όλη αυτή την πρόοδο σε παγκόσμιο επίπεδο και αυτό είναι το ε, συμπέρασμά μου. Πέραν της καινοτομία και των νέου ορίζοντα αυτού του ανοιχτού πεδίου του διαστήματος, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να είναι ηγετική δύναμη ε, στα διαστημικά συστήματα, το είδαμε με τον, με τον έχει τεχνολογικούς ε, φορείς και επιχειρήσεις ε, πολύ καινοτόμους, αλλά έχει να αντιμετωπίσει τις ρήξεις και τις προκλήσεις όχι μόνο των ε, χωρών των αναπτυσσομένων στο διάστημα, αλλά κυρίως τον ανταγωνισμό των παραδοσιακών ισχυρών δυνάμεων. όλα αυτά θα χρειαζόντουσαν μια εξαντλητική μελέτη, αλλά ας πούμε ότι θα πρέπει να έχουμε συνείδηση όχι μόνο της ε, παρακολούθησης του επίπεδου του διαστήματος, αλλά της υποστήριξης ε, των αμυντικών μας ε, επιχειρήσεων για να μην βρεθούμε σε ένα διπλό αρνητικό σενάριο που αφενός θα μέναμε πίσω από τις πρώτες χώρες ε, Ρωσία, Ηνωμένε Πολιτείε, Ινδία και Κίνα αλλά θα μπορούσαν και να μας φτάσουν οι χώρες που αυτή τη στιγμή προχωρούν στο διάστημα. Απομάκρυνση λοιπόν από τους ε, πρώτους και πλησίασμα από τους τρίτους αν θέλετε. Και η διαστημική μας στρατηγική αυτή τη στιγμή προσπαθεί να αποτρέψει και τα δύο αυτά δεν μπορούμε να χάσουμε τον ανταγωνισμό ε, στο πεδίο του διαστήματος όπως είχαν δηλώσει και η ηγεσία της ε, γαλλικής αεροπορίας πρόκειται για μια κρίσιμη στιγμή χρειάζεται ένα άλμα και μια κοινή προσπάθεια μια σύγκληση προσπαθειών κάθε κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αμυντική προσπάθεια του διαστήματος με θέληση συνεργασίας με τους διεθνείς φορεί φορείς ώστε να οικοδομήσουμε ένα πεδίο ειρήνης στο διάστημα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες αυτές. Δίνω το λόγο στον Πασκάλ Κλοντέλ. Είστε Chief Operating Officer της GSA, η οποία δημιουργήθηκε λόγω της στρατηγικής σπουδαιότητας των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ε, ε, ε, ε, ε δορυφορικής και θα θέλαμε να υπάρξει υποστήριξη για τον τομέα αυτόν. Η JSA θα αναλάβει νέες αποστολές δεδομένου του νέου κανονισμού για το διάστημα. Κύριε Κλοντέλ, είστε έμπειρο γνώμων στον τομέα του διαστήματος. Έχετε εμπειρία πάνω από 30 χρόνια. Θα μπορέσετε να μας διαφωτίσετε για την επιχειρησιακή υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Προγράμματος και για τις διαστημικές δυνατότητες άμυνας και ασφάλειας της Ευρώπης με στόχο την προστασία των δικών μας υποδομών. Τα διαστημικά μας μέσα έχουν στρατηγική σπουδαιότητα σε θέματα μη στρατιωτικά, στρατιωτικά, εμπορικά, άμυνας και ασφάλειας και θα πρέπει να διασφαλίζουν ευρωπαϊκή πρόσβαση στο διάστημα ανεξάρτητη με δυνατότητα προστασίας των υποδομών μας και ειδικότερα από τα διαστημικά απόβλητα. Σας δίνω το λόγο για το πολύ 10 λεπτά για να δώσουμε μετά το λόγο ε, να περάσουμε σε μια φάση πιο διαδραστική αργότερα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ε, αγαπητοί βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι, να σας ευχαριστώ που μου δίνετε σήμερα την ευκαιρία να σας παρουσιάσω τα διαστημικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την τεχνογνωσία μας. Μας βοηθούν να έχουμε στρατηγική αυτονομία ως Ευρωπαϊκή Ένωση και να ενισχύσουμε την πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Πράγματι, τα διαστημικά προγράμματα προσφέρουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση βασικά εργαλεία για την αυτονομία στην λήψη αποφάσεων μέσω των υπηρεσιών ε, πλοήγησης, γεωσκόπησης, ε, ε, τηλεπικοινωνιών και επιτήρησης. Να σας υπενθυμίσω στον πόλεμο του κόλπου, είχαμε το παράδειγμα των ε, δορυφόρων ε, γεωσκόψης που μας επέλεξαν να κάνουμε άλλες επιλογές από τη Αμερικανή. Όπως ξέρετε η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μοναδική διότι ανέπτυξε με μη στρατιωτική προσέγγιση τα διαστημικά συστήματα ε, διασφαλίζοντας και τα κρατικά συμφέροντα. Αυτό το ονομάζουμε διτό χαρακτήρα. Το Ταμείο σήμερα έρχεται να ενισχύσει Όλε αυτέ τι δυνατότητε που διαθέτουν τα κράτη-μέλη και ενισχύει του δεσμού μεταξύ διαστήματο, άμυνας και ασφάλεια. Μην ξεχνάμε λοιπόν ότι, είπατε, ο νέο κανονισμό που ψηφίστηκε τον περασμένο Απρίλιο ενισχύει αναμφίβολα το δεσμό αυτό μεταξύ διαστήματο άμυνας και ασφάλεια και δημιουργεί συνέργειε μεταξύ προγραμμάτων πλοήγησης, γεωσκόψης τηλεπικοινωνιών. Αυτές οι συνέργειες ε, πράγματι βελτιώνουν τα εργαλεία, τις εφαρμογές όπως για παράδειγμα την ανείχνευση και την καταπολέμηση φυσικών καταστροφών, τη μετανάστευση, την θαλάσσια επιτήρηση των ανοιχτών των συνόρων. Σε αυτά, όπως είπατε, πρέπει να προσθέσουμε την ανάπτυξη της επιτήρησης του διαστήματος με το πρόγραμμα Space Situational Awareness, πολύ βασικό για να διασφαλίσετε η προστασία των διαστημικών μας μέσων. Ειδικότερα μετά από τις δοκιμές, αντιδορυφορικές δοκιμές που ανέφερε ο συνάδελφος. να σας παρουσιάσω την αποστολή της GSA. Είναι ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιφορτισμένος με τα ε, προγράμματα ε, δορυφορικής πλοήγησης. Το Galileo είναι ένας ε, οργανισμός επιχειρησιακός της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιφορτισμένος με τη λειτουργία των συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης και την παροχή υπηρεσιών για να διασφαλίζει την ασφάλεια στο επίπεδο επιχειρήσεων και υπηρεσιών και για την πρόθεση της χρήσης τους των ε, υπηρεσιών Galileo και Έγνος σε όλου του τομεί τη οικονομίας. Αυτό που ονομάζουμε New Space. Αυτέ οι υπηρεσίε Galileo έγνωση είναι προσπελάσιμε για του μη στρατιωτικού επαγγελματίε, θεσμικούς και κυβερνητικού ε, χρήστε. Όπω καταλάβατε η ασφάλεια δεν είναι παρά ένα από του τρει πυλώνε τη GSA. Περιλαμβάνει και το Συμβούλιο Εγκριση τη Ασφάλεια, το ΣΑΒ, όπω ονομάζεται αυτό, είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμό που υποστηρίζεται από τον οργανισμό μα και διασφαλίζει τη συμμόρφωση των προγραμμάτων Γαλιλαίο και Έγκνο με τους κανόνε ασφάλεια ε, της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Το Γαλιλαίο λοιπόν σχεδιάστηκε για να διασφαλίζει την αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ε, δορυφορικής πλοήγησης. Αυτό είναι το Γαλιλαίο. Τι είναι ακριβώς, ε, βασίστε σε μια περίπλοκη υποδομή για να παρέχει ένα σήμα πολύ μεγάλη ακρίβεια. Σήμερα η ακρίβεια που έχει είναι καλύτερη από αυτή των τεσσάρων μεγάλων υπαρχόντων συστημάτων. Το σύστημα είναι περίπλοκο λόγω του χρονικού συγχρονισμού σε ε, εκατομμυριωστό του δευτερολέπτου για να παρέχει υπηρεσίε ε, ακρίβεια θέση και χρόνου και περίπλοκο επίση, όσον αφορά τη διαχείριση των 22 δορυφόρων που λειτουργούν για, από πλευρά Ευρώπη αποτελείται από ένα διαστημικό σκέλο και ένα επίγειο σκέλο. Το διαστημικό σκέλο, όπω ξέρετε, αποτελείται από δορυφόρου και από εκτοξευτήρες ε, το επίγειο σκέλος ε, έχει όλα τα συστήματα διαχείρισης ε, που διαχειρίζονται τους δορυφόρους και τις πληροφορίες που έρχονται από αυτούς. Βασίζονται σε 200 ελέγχους, 200 κέντρα ελέγχους στην Ιταλία και στη Γερμανία. Τον Καλήλιο επίσης βασίζεται σε δύο κέντρα ασφα... επιτρήσης ασφάλειας, τα GSC, που παρακολουθούν 24 ώρες το 24 ώρες, 7 ημέρες τη βδομάδα, το... σε επίγειες εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες. Τρει ε, υπηρεσίε ε, παρέχει το Γαλιλαίο από το Δεκέμβριο του 2017. Το Open Service που γνωρίζετε όλοι θα έχετε στο smartphone σα με μεγάλη ακρίβεια πάνω από ένα δισεκατομμύριο Χρήστε μέχρι σήμερα. Το Search and Rescue που είναι η υπηρεσία έρευνα και διάσωση. επιτρέπει τον εντοπισμό ανθρώπων που κινδυνεύουν το 10 λεπτά μέχρι την ανείχνευση με ακρίβεια και χιλιόμετρου σε σχέση με τα 45 λεπτά που είχαμε παλιότερα και την ακρίβεια των 5 χιλιόμετρων που είχαμε χωρί το Γαλιλαίο και μετά έχουμε το PRS, Public Regulated Service, δημόσια ρυθμισμένη υπηρεσία που αφορά ειδικά τις ε, κρατικές αποστολές. Τώρα θα σας παρουσιάσω τρία σημεία ιδιαίτερα, το PRS, ε, τις κρίσιμες υποδομές και την ασφάλεια. Αυτοί οι τρεις τομείς ε, είναι τομεί με του οποίου έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία η GSA. Αυτή την εμπειρία θα τη διαθέσει σε όλα τα διαστημικά προγράμματα μέσω του νέου κανονισμού. Δεδομένου ότι η GSA θα έχει διευρυμένο αντικείμενο μετά από την 1η Ιανουαρίου του 2021 το PRS είναι ο ακριβωνιός λήθης της χρήσης των διαστημικών προγραμμάτων στην Ευρώπη. Ε, παίζει θεμελιώδη ρόλο, δημιουργεί μια λυσίδα ασφάλεια μέσω κρυπτογράφηση προσαρμοσμένη στι ανάγκε των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτρέπει ε, την κοινή χρήση κονδυλίων για δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η σταθερότητα και η αξιοπιστία του συστήματο αυτού δορυφορική πλοήγηση είναι αναγκαία. Αυτό συνεπάγεται συνέχεια, ε, απαιτεί συνέχεια των ε, υπηρεσιών, αποτελεσματική λειτουργία και ασφάλεια υψηλού επίπεδου για την προστασία όλων των υποδομών και των επικοινωνιών μέχρι τον τελικό χρήστη. Η εμπειρία αυτή που έχουμε αποκτήσει για το PRS παίζει σημαντικό ρόλο για την κοινή χρήση των μέσων πλοήγησης Γαλιλαίου, τηλεπικοινωνίας δορυφορικών επικοινωνιών και διαστημικής επιτήρησης, δεδομένου ότι το βήμα αυτό της αγοράς ε, είναι ουσιαστικά τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να επιστήσω τώρα την προσοχή σας ε, στην προστασία των κρίσιμων υποδομών στην Ευρώπη και στο συγχρονισμό με τα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης. Ο συγχρονισμός αυτός σήμερα διασφαλίζεται από το σύστημα GPS, το, το αμερικανικό Γαλιλαίο. Είναι σημαντικό λοιπόν η νομοθεσία να προωθήσει το Γαλιλαίο ως κύριο προμηθευτή υπηρεσιών ώστε να είμαστε ανεξάρτητοι όσον αφορά αυτές τις κρίσιμες υποδομές στην Ευρώπη. Η προσθέμενη αξία τη ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική σε θέματα εσωτερική ασφάλεια είναι λοιπόν πολύ σημαντική. Μπορούμε να ε, επηρεάσουμε έτσι τις ε, ε, μεταφορές, στην ενέργεια, την ασφάλεια και τις τράπεζες. Και τέλος, όσον αφορά την ασφάλεια, για να ενισχύσουμε την πολιτική ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρειάζεται η συμβολή των δορυφορικών μέσων. Οι διαστημικές δυνατότητες πρέπει να περιλαμβάνουν και την έννοια της ασφάλειας από σχεδιασμού, ώστε να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις απειλές και τις αδυναμίες των συστημάτων. Πόσο μάλλον που Απειλέ εξελίσσονται διαρκώς ε, για τις υπηρεσίες μας και εντείνονται τα τελευταία χρόνια. Έτσι οι μηχανισμοί προστασίας πρέπει να είναι πιο ευέλικτοι και να προβλέπουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις εξέλιξει αυτέ. Μέσω του Γαλιλαίου σε θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο έχουμε ε, σημαντική κοινή χρήση των διαστημικών πόρων ε, που εξυπηρετούν τις πολιτικές ασφάλειας και άμυνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον ε, η εμπειρία του ΣΑΡ, του Συμβουλίου Έγκρισης της Ασφάλειας, ε, είναι πολύ σημαντική για την προστασία των διαστημικών μας ε, υπηρεσιών και των σχετικών υπηρεσιών. Πριν κλείσω, θα ήθελα να επιμείνω στην στρατηγική διάσταση του διαστήματος. Είναι σημαντικό να διατηρήσουμε τις τεχνολογικές και βιομηχανικές δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό απαιτεί παρουσία στη μη στρατιωτική αγορά. Αυτό θα κάνει μεγάλη διαφορά και σε θέματα δημοσιονομικά σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας. Γι' αυτό τον <coughs> λόγο ε, έχει ως αποστολή ο οργανισμός μας τη χρήση συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης, τα αγκαλιλαίου και τα Έγνος και θέλει να τα χρησιμοποιήσει όλους τους κλάδους αγοράς του New Space ε, διασφαλίζοντας έτσι ε, ε, και το μέλλον των βιομηχανιών μας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μας. Επιτρέπει επίσης την δημιουργία λύσεων ε, καινοτόμων και ανταγωνιστικών για να έχουμε μια βιομηχανία ακόμα πιο ανταγωνιστική στη διεθνή αγορά. Και επίσης επιτρέπει η οικονομική ανάπτυξη σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να κλείσουμε, θα ήθελα να υπογραμμίσω και πάλι το γεγονός ότι οι διαστημικές υποδομές ε, είναι υψηλού επίπεδο, το ίδιο και η τεχνογνωσία μα και με υψηλέ επιδόσει. Έτσι, έχουμε το απαραίτητο το που απαιτείται για να ηγηθούμε σε θέματα πολιτική ασφάλεια και άμυνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον ε, κύριο Κλοντέλ, ευχαριστούμε που τηρήσατε και το όριο χρόνου. Κυρία Καρίν Κλέης, είσαστε ειδική απεσταλμένη της ΙΕΔ από τον Ιούλιο του από τον Ιούλιο φέτος και ήσασταν υπεύθυνοι της Task Force ε, για τα διαστημικά μέσα τα ευρωπαϊκά από το 2005. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την διαθεσιμότητά σας σήμερα να συμμετάσχετε σε αυτήν την ε, συζήτηση, σε αυτήν την ακρόαση. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τις πρωτοβουλίες σας ε, και πώς συμπεριλαμβάνετε τη διαστημική διάσταση στην κοινή πολιτική ασφαλείας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μας μιλήσετε και για μια ε, διπλωματική πρωτοβουλία ώστε να έχουμε μια βιώσιμη και υπεύθυνη ε, εξωτερική δράση, τα τρία σως που λέμε και ίσως ε, νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα μπορούσαμε να λάβουμε στο κατάλληλο επίπεδο εθνικό ή υπερεθνικό. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε να έρθω στην Επιτροπή σας σήμερα. Είναι υπο-επιτροπή, αν και για μένα το έργο της είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα έπρεπε ίσως να είναι κανονική επιτροπή. Θα ήθελα να ξεκινήσω με μια πολύ σύντομη παρουσίαση των αρμοδιοτήτων της υπα της εκπροσώπου και του επιτελείου της ε, καθώς και της ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης στον χώρο του διαστήματος. Όπως είπε η Επίτροπος Μπιενκόφσκα, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης είναι το Υπουργείο Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τροποντινά. Γνωρίζουμε πώς δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη διατύπωση, όμως στην πράξη αυτό κάνουμε. Η, η πατή εκπρόσωπος έχει δύο κύριες αρμοδιότητες σε ό,τι αφορά το διάστημα. Καταρχάς, η απόφαση του Συμβουλίου 496 του 2014 δίνει στον υπατό εκπρόσωπο και στο Συμβούλιο αρκετά μεγάλες ευθύνες στην αντιμετώπιση απειλών. Απειλών για το παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης, είτε το Γκαλιλαίο είτε το Έγνος. Έχουν προβλεφθεί λοιπόν οι κατάλληλε διαδικασίες έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε και να ασκήσουμε τα καθήκοντά μας σε περίπτωση απειλής. Έπειτα, η δεύτερη αρμοδιότητα είναι η διεύθυνση του δορυφορικού κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, το οποίο είναι μια μοναδική ικανότητα στην Ευρώπη για συλλογή πληροφοριών από το διάστημα. Υπάρχουν και πρόσθετες αρμοδιότητες σε ό,τι αφορά το διάστημα διάφορες διπλωματικές δράσεις στο πλαίσιο της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης, συμμετοχή σε πολυμερή φόρα όπως τα Ηνωμένα Έθνη, ε, όπου συμμετέχουμε μαζί με τα κράτη-μέλη και δημόσια διπλωματία. Θα επανέλθω πάνω σε αυτό. Επίσης, λειτουργούμε συμβουλευτικά προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του ρόλου του, του εκπροσώπου ως Αντιπρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πρόεδρου του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων και επικεφαλής της, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει κομβικό ρόλο σε θέματα ασφάλειας και άμυνας, βρίσκεται στο κέντρο συνεργασίας μεταξύ Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ε, υπόλοιπων σχετικών οργανισμών. με στόχο την εφαρμογή της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την αυτονομία της και τη δημιουργία συνεργειών. Θεωρώ επομένως ότι ο ρόλος του ΙΠΑ του εκπρόσωπου είναι πάρα πολύ σημαντικός ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το θέμα της σημερινή μας ακρόασης. Το διάστημα είχε από πολύ νωρί στρατιωτικό χαρακτήρα. Το Μάρτιο του 1954 εκδόθηκε η έκθεση RAND μέσα στον ψυχρό πόλεμο, η οποία προέβλεπε ένα σύστημα δορυφορικής αναγνώρισης ε, και το χαρακτήριζε ως στρατηγική σημασίας για την Ευρώπη. Τότε μπήκαν τα θεμέλια της ε, διαστημικής βιομηχανίας. το διάστημα έχει κυρίω στρατιωτικό χαρακτήρα για πολλέ χώρες, ακόμα και σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει όμω υιοθετήσει εκ διαμέτρου αντίθετη στάση, δημιουργώντα διάφορα προγράμματα πολιτικού χαρακτήρα, με τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν και στρατιωτικά. Όμως τα προγράμματα και τα συστήματα αυτά έχουν ε, δημιουργηθεί για πολιτικούς σκοπούς. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που περιλαμβάνονται σε, αυτόν τον, ε, σε αυτά τα προγράμματα πολιτικού χαρακτήρα. Αλλά το 1967 υπογράφει και ετέθη σε ισχύ η συνθήκη για το διάστημα και άλλα νομικά κείμενα των Ηνωμένων Εθνών, κείμενα πάρα πολύ σημαντικά έτσι ώστε να παραμείνει ειρηνική η χρήση του διαστήματος στον κόσμο. Οι βασικές λοιπόν αρχές ε, είχαν να κάνουν με την διερεύνηση και εξερεύνηση του διαστήματος ε, για το καλό της ανθρωπότητας, καμία κυριαρχία από μία μόνο χώρα, διατήρηση της ε, ειρήνης και χρήση του διαστήματος για ειρηνικούς σκοπούς, χωρίς πυρηνικά, χωρίς πυρηνικές δοκιμές ή δοκιμές οποιονδήποτε άλλων όπλικων συστημάτων ή στρατιωτικών επιχειρήσεων. Σήμερα που βρισκόμαστε, η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας έχει επιπτώσεις και στο διάστημα. Το 60% της οικονομίας εξαρτάται έμεσα ή άμεσα από διάφορα εργαλεία που χρησιμοποιούν ε, το διάστημα. Υπάρχει η τεχνητή νοημοσύνη και το διαδίκτυο των πραγμάτων και δίχως αμφιβολία το διάστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πάρα πολλούς ε, τρόπους και έχει τεράστιο δυναμικό. Αυτό βέβαια μας καθιστά και ευάλωτους σε θέματα προστασίας των διαστημικών μας υποδομών. Ο κύριος ε, Ζάζετς είπε ότι την περίοδο του ψυχρού πολέμου ε, είχαμε ένα δίπολο, όμως ε, τώρα έχουν, ε, έχουν αναδυθεί αρκετές υπερδυνάμεις, υπάρχουν πολλοί πόλοι ισχύς και νέοι παίκτες στο διάστημα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να τα αναγνωρίσουμε αυτό, καθώς επίσης και τον ορισμό του νέου διαστήματος, κάτι που αρνείται η Ρωσική Ομοσπονδία, διότι το θεωρεί αντίθετο στην συνθήκη του 1967. Η συνθήκη του 1967 προβλέπει ότι τα κράτη έχουν συλλογική διεθνή ευθύνη για τις πράξεις τους, έστω και αν αυτές γίνεται από ένα μονομένο κράτος. Τώρα, το περιβάλλον στο διάστημα χαρακτηρίζεται από λεώνα και περισσότερη συμφόρηση και ανταγωνισμό. Υπάρχουν πολλά σκάφη, υπάρχουν πολλά υπολείμματα που βρίσκονται σε τροχιά. Πάνω από 20.000 υπολείμματα σκαφών αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε τροχιά και δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν τον αριθμό τα υπολείμματα που έχουν ε, διαστάσεις μικρότερες του 1 εκατοστού. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει τον ε, την Αμερικανική Αστρονομική Κοινότητα να αναφερθεί στις ε, αρνητικές επιπτώσεις. Με άλλα λόγια, στο φαινόμενο Κέσλερ. Όταν δηλαδή η υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση σωματιδίων στο διάστημα, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για ε, σύγκρουση με αρνητικές επιπτώσεις για ε, τις επόμενες γενιές. Βλέπουμε όμως ότι σε μια εποχή που η οικονομία μας εξαρτάται στο 60% από διάφορες διαστημικές εφαρμογές, είναι σχεδόν αδύνατο να μην χρησιμοποιήσουμε το διάστημα και να μην αναγνωρίσουμε λοιπόν ε, τα προβλήματα αυτά υπάρχουν διάφορες απειλές, ε, jamming, spoofing, ε, κυβέρνο απειλές, κινητικές απειλές, ASAT και διάφορες απειλές που έχουν να κάνουν με τον ανταγωνισμό, δηλαδή με το γνωρισμό του νέου διαστήματος ή με τις νέες δυνάμεις που χρησιμοποιούν το διάστημα για να εκφράσουν την ισχύ τους. Όπως έχουμε ήδη συζητήσει στο παρελθόν. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε και ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν. Ας επικεντρωθούμε λίγο στην ε, δράση της, είπα, εκπροσώπου και της ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ε, η υπηρεσία αυτή, βοηθούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, αλλά και τα κράτη-μέλη, έχουν αρκετέ δυνατότητες. Υπάρχουν παράλληλες αρμοδιότητες στο διάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 4 και το άρθρο 189 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε ήδη ότι υπάρχουν τρία κύρια στοιχεία. Υπάρχει η δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε τις αρμοδιότητες τύπτας εκπροσώπου έτσι ώστε να προωθήσουμε την ασφάλεια στο διάστημα και να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση των ε, διαφόρων μέσων που διαθέτουμε. Επίσης, αναφέρθηκα ήδη στον κανονισμό του 2014, τον 496, όπου αναφέρεται ο οποίος αναφέρεται στην επιχειρησιακή αλυσίδα ασφάλειας του συστήματος Γκαλιλαίου. Η Υπηρεσία λοιπόν στατική Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρμόδια και για την επιχειρησιακή αλυσίδα ασφαλεία. Επίσης, το δορυφορικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τις αρμοδιότητές μας, όμως υπάρχουν αρκετές προκλήσεις, ε, υπάρχει υποχρηματοδότηση αυτή τη στιγμή, χρειάζεται λοιπόν μια αύξηση της χρηματοδότησης έτσι να ώστε να μπορέσει να γίνει πλήρως λειτουργικό. Εν ώψη του νέου πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου, λοιπόν, θα χρειαστεί να γίνουν κάποιε προσαρμογέ έτσι ώστε η δυνατότητα συλλογική και επεξεργασία πληροφοριών τη Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί αυτόνομη. Τι προτείνουμε, λοιπόν, να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού 496 ώστε να περιλαμβάνει όλα τα στατικά στοιχεία του διαστημικού προγράμματο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το μέλλον, εφόσον και όταν αυτό εγκριθεί. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει συμφωνία επί της ουσίας από τον νομοθέτη, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο δηλαδή για τον κανονισμό και μόνο το Συμβούλιο για την απόφαση και με το που διαλευκανθούν όλα τα, ε, τα οριζόντια σημεία θα εξεταστεί ξανά η Επίσης, υπάρχει και η πρωτοβουλία της δημόσιας διπλωματίας, τα τρία σως, όπως είπε και η Πρόεδρος. Είναι μια έκκληση για υπεύθυνη συμπεριφορά και για βιώσιμη χρήση του διαστήματος, για την δημιουργία ενός κώδικα διαντολογίας για ε, προς των μελλοντικών γενναίων. Γιατί τρία σως, γιατί είναι τα τρία S, security, safety και sustainability, δηλαδή ασφάλεια και αηφορία. Αλλά και τρία σώσε διότι το, ο χαρακτήρας είναι επίγον. Η πρόθεση αυτής της ε, πρωτοβουλίας μας είναι να συνεργαστούμε με εσάς, ε, τους ε, πολιτικούς, του υπεύθυνου λήψη αποφάσεων, την ε, κοινωνία των πολιτών, τη βιομηχανία, την πανεπιστημιακή κοινότητα και τους διαστημικούς οργανισμούς σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε να προωθήσουμε την ε, βιώσιμη και υπεύθυνη συμπεριφορά στο διάστημα. Όπως ε, λοιπόν και τις δεκαετίες του 1950 και του 1960 θα πρέπει και τώρα να τεθούν κάποιοι κανόνες για το διάστημα έτσι ώστε να αποφύγουμε τις διστάρεστες συνέπειες και τις συγκρούσεις. Αυτό σημαίνει ότι κάθε εκτόξευση δορυφόρου θα πρέπει να έχει γίνει μελετημένα και να προβλέπεται η απόσυρσή του στο τέλος ε, της ε, διάρκειας ζωής του. Ε, ενδεχομένως επίσης μία διαχείριση της κίνησης στο διάστημα με αναμεταδότες όπως ε, συμβαίνει στο IFF ή όπως συμβαίνει στη θάλασσα. Φυσικά δεν είναι ρόλος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης να ορίσει τα μέτρα, όμως μπορούμε να κάνουμε προτάσεις για τους ε, ειδικού. Αυτό που εμείς επιθυμούμε είναι να οδηγηθούμε σε συνένεση έτσι ώστε να υπάρξει υπεύθυνη διαχείριση του διαστήματος από όλους τους φορείς. Και εδώ φτάνω στον τέταρτο άξονα δράσης για ε, την Υπηρεσία εξωτερική δράση και την Υπατή Εκπρόσωπο, δηλαδή να δημιουργήσουμε κάποιο εθελοντικό όργανο εντό τη Ένωση και των κρατών μελών, το οποίο θα οδηγήσει σε νομικά δεσμευτικές αποφάσεις μακροπρόθεσμα. Αυτό το εθελοντικό όργανο φυσικά θα προωθήσει τις κοινέ δηλώσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών, θα συμμετέχει στα διεθνή φόρα και στα Ηνωμένα Έθνη και θα κάνει έκκληση για υπεύθυνη συμπεριφορά. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να συνεργαστούμε για μια ηθική, ασφαλή και βιώσιμη χρήση του διαστήματος. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στην κυρία Σιμονέτα Διπίπο που είναι διευθύντρια του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών της ε, ε, θεμάτων του εξώτερου διαστήματος. Επίσης ε, είστε υπεύθυνοι του UN Spider που είναι μια πλατφόρμα αντιμετώπισης κρίσεων και καταστροφών. Ο Γενικός Γραμματέας σας έχει αναθέσει ε, τα θέματα της ειρηνικής χρήσης της διαστημικής τεχνολογίας. Είχα διαβάσει και ότι ένας αστεροειδής, ο 21887, φέρει το όνομά σας τιμώντας ε, τη συνεισφορά σας στο, στα θέματα του διαστήματος. Επίσης να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που έχουμε μια ισορροπία φίλου σε αυτό το πάνελ. Δεν μας συμβαίνει πάρα πολύ συχνά σε θέματα αμήνης και ασφάλειας. Μακάρι να μπορούσαμε πιο συχνά. Τώρα, με την ε, αύξηση της ε, ανθρώπινης χρήσης στο διάστημα, της τεχνολογίας, των μέσων, Χρειαζόμαστε μια χρηστή διαχείριση των πόρων. Ε, θα μας αναφέρετε τις ε, βασικότερες γραμμές της βιωσιμότητας ε, της διαχείρισης αυτής, όπως θα μας αφέρετε και την εξέλιξη των εργασιών στο ΚΟΠΟΥΟΣ, την Επιτροπή για την Ειρηνική Χρήση του Εξωτερικού Διαστήματος, Επίσης, τι περιμένετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να ενισχυθούν αυτέ οι κατευθυντήριε γραμμέ και η ειρηνική χρήση του διαστήματο. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ και για την εξαιρετική αυτή εισαγωγή που κάνατε, αξιότιμα μέλη Ω υπεύθυνη του Γραφείου των Ηνωμένων Αθηνών για τα θέματα του διαστήματος είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα να είμαι εδώ μπροστά σα, εκπροσωπώντα τα Ηνωμένα Έθνη. Τα Ηνωμένα Έθνη και το Γραφείο των ε, Θεμάτων Εξώτερου Διαστήματος, του UNOSA, είναι μια ε, ευκαιρία ε, εξέτασης των δραστηριοτήτων στο διάστημα, της επιστήμης, της τεχνολογίας αλλά και του νομικού πλαισίου. Κατέχουμε λοιπόν μια στρατηγική θέση εντός της δομής των Ηνωμένων Εθνών ως προς την ενίσχυση του δυναμικού των μέσων για το διάστημα. Τώρα, η πρόσβαση στο περιβάλλον του διαστημικό ε, και η χρήση των σχετικών μέσων είναι πιο σημαντική παρά ποτέ. Είχαμε 60 νέους δορυφόρους με ενιαία εκτόξευση. Έχουμε πάρα πολλά ε, ε, σώματα σε τροχιά εκτός από δορυφόρους και άλλα συστήματα και εκτός από τους χιλιάδες αυτούς δορυφόρους και άλλα μέσα που βρίσκονται σε τροχιά πρέπει να αναπτύξουμε μια κοινή κατανόηση του τι σημαίνει μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της διαστημικής δραστηριότητας. Και αυτό είναι ο... Και είναι πολύ ενθαρρυντικό μάλλον να βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να προσπαθεί να αντιμετωπίσει κάποιες από τις πιο επίγουσες προκλήσεις που έχουμε σήμερα πρέπει να εστιαστούμε στις ανισότητες, στη φτώχεια, στις ε, δημογραφικές τάσεις, ε, στην κλιματική αλλαγή, στις κρίσεις, στην τεχνολογική ε, καινοτομία που χρειάζεται για να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Οι προκλήσει αυτέ πρέπει να αντιμετωπιστούν και από το ΗΕ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε λοιπόν να συνεργαστούμε και ελπίζω πράγματι να βρούμε έναν τρόπο να συνεργαζόμαστε περισσότερο, πιο στενά, στην αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών. Το πρόγραμμα UN Spider αναφέρθηκε. Εμείς ε, διαχειριζόμαστε το πρόγραμμα αυτό από το 2006. Μιλούμε για την ε, πλατφόρμα των Ηνωμένων Εθνών για την αντιμετώπιση επιγουσών αναγκών και κρίσεων και μιλούμε για τα 193 μέλη, κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με διαστημική δυνατότητα απεικόνησης και άλλων τεχνολογικών υπηρεσιών ώστε όλα τα κράτη να μπορούν να εκμεταλλευτούν ε, το δυναμικό αντιμετώπισης ε, καταστροφών και κρίσεων μέσω της διαστημικής τεχνολογίας και της άμεσης ανταποκρίσης. Επίσης έχουμε ένα άλλο πρόγραμμα εδώ και 15 χρόνια, το ICG, Διεθνής Επιτροπή στα Δορυφορικά Συστήματα Πλοήγησης, όπου έχουμε τους τέσσερις βασικούς παρόχους τους Κινέζους, τους Ευρωπαίους με την GNSS, ε, έγνωσκε και Γαλιλαίο, τους Αμερικανούς με το GPS και τους Ρώσους με τον Κλώνας. Αυτά, αυτός μάλλον είναι ένας τρόπος ε, διαλειτουργικότητας για το πλαίσιο, για το σύστημα αυτό και για παροχή υπηρεσιών παντού στον κόσμο. Τώρα πρόσφατα πέρυσι είχαμε ε, αναθέσει μία μελέτη μαζί με την GSA, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό, ε, συνδυάσαμε το Κοπέρνικος και το EEGNSS και 169 στόχους που είναι υπό τους 17 ε, στόχους βιωσίμου ανάπτυξης που είναι στόχοι όπως γνωρίζετε για όλα τα κράτη-μέλη μέχρι το 2030 ευρύτατη και επί διαφόρων θεματικών. Βρήκαμε λοιπόν, αναλύοντας τον καθέναν από τους στόχους αυτού, ότι το 40% εξ αυτών εξαρτώνται από την παρατήρηση της γης από δορυφορικά στήματα. Και αν, προσθέσουμε και τις τηλεπικοινωνίες, εκτιμούμε ότι το ποσοστό αυτό θα ήταν άνω το 60%. Δηλαδή κανείς στον κόσμο δεν μπορεί να κάνει τίποτε στην πραγματικότητα χωρίς διαστημική τεχνολογία. Και παρά τους βιώσιμους στόχους, χρειαζόμαστε και περισσότερες ευκαιρίες για την πρόσβαση στο διάστημα. Το 2018 προχωρήσαμε μια πρωτοβουλία που ονομάζεται πρόσβαση στο διάστημα για όλους για την οικοδόμηση εταιρικών σχέσεων σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα ώστε να βοηθήσουμε περισσότερες χώρες να έχουν πρόσβαση στο διάστημα για ερευνητικές και δορυφορικές δραστηριότητες με βιώσιμο και υπεύθυνο τρόπο. Δεν φέρνουμε νέους παίκτες στο διαστημικό πεδίο χωρίς να τους υποστηρίξουμε χωρίς να τους παρέχουμε ένα πλαίσιο υπευθυνότητος. Έχουμε λοιπόν συνεργάτες από τον ιδιωτικό τομέα που σας έλεγα. Μαζί με την Airbus είχαμε προχωρήσει σε ένα πρόσφατο πρόγραμμα να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη στην δική τους πλατφόρμα τη διαστημική. Έχουμε επίσης με την Κινέζικη Διαστημική Υπηρεσία μια συνεργασία και επιλέξαμε πρόσφατα εννέα πειραματικές δοκιμές στον ε, διαστημικό σταθμό της Κίνας. Εννέα περιπτώσεις που επιλέχθηκαν από όλο τον κόσμο, από όλο τον πλανήτη, με επιστημονική αξία. Έχουμε και με την ESA, με ερευνητικά κέντρα συνεργασία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με ευρωπαϊκές εταιρείες. Και πέρυσι ήταν πολύ ενδιαφέρον όταν μέσω συμφωνίας με την ε, ε, η Ιαπωνική Υπηρεσία Διαστημικής Έρευνας καταφέραμε μια χώρα να εκτοξεύσει τον πρώτο δορυφόρο, αυτή ήταν η Κένια. Για πρώτη φορά ε, κατάφεραν να εκτοξεύσουν δορυφόρο. Αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με Γουατεμάλα, Ινδονησία, Μαυρίκιο, Μολδαβία και άλλους που έχουν επιλεγεί για την προετοιμασία. Υποστηρίξαμε λοιπόν την Κένια να αναπτύξει ένα διαστημικό νομικό πλαίσιο και μια υπηρεσία ώστε να μπορέσει να ρυθμίσει αλλά και να εγγράψει τη δραστηριότητα της αυτή στο πλαίσιο των ΗΠΑ. Και έχουμε την υπηρεσία της, ε, των ΗΠΑ για την ειρηνευτική χρήση του εξώτερου διαστήματος. Έχουμε διάφορες οντότητες όμως που είναι ε, συνδεμένες μεταξύ τους το πλαίσιο αυτό είναι πολύ χρήσιμο για την ανάπτυξη ενός διεθνούς νομικού πλαισίου και είναι το βασικό διακυβερνητικό βήμα για την συνεργασία και την υπεύθυνη έρευνα και χρήση του διαστήματος. Η UNOSA, που είναι ο μόνος φορέας που αφιερώνεται 100% στα διαστημικά θέματα στα Ηνωμένα Έθνη, έχει ένα ρόλο πολύ ευρύ. Είμαστε, αν θέλετε, κάτι σαν παγκόσμιος διευκολυντής, πλατφόρμα, ερχόμαστε σε επαφή για να αναπτύξουμε το δυναμικό, για να βελτιώσουμε τις δεξιότητες και τη γνώση όλων των ε, ενδιαφερομένων φορέων. Βοηθούμε τα κράτη-μέλη να συστήσουν νομικά και ρυθμιστικά πλαίσια για να ε, διακυβερνήσουν τη διαστημική τους δραστηριότητα και να ενισχύσουν την ικανότητα της υπεύθυνης χρήσης ε, των χωρών του χώρου του διαστήματος και η ΟΝΟΣΑ και η Κόπιος ε, ήταν κεντρική σημασία για την εφαρμογή και υπογραφή συμφωνιών ώστε να διατηρήσουμε ε, το διάστημα ως χώρο ανθρώπινης συνεργασίας και ώστε να έχουμε ε, ένα ασφαλές διάστημα και βιώσιμο διάστημα μέσω μιας παγκόσμιας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τις δραστηριότητες αυτές έχουμε τον, το Μητρό των Ηνωμένων Αθνών και τις βιώσιμε κατευθυντήριες γραμμές διαφάνειας και ανάπτυξης ε, μέσων εμπιστοσύνης. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικές περιοχές στην εργασία που εστιάζονται στην πιο υπεύθυνη και βιώσιμη στάση που πρέπει να έχουν οι χώρες ε, στο διάστημα και για τις οικονομικές τους και εμπορικές δραστηριότητες το μητρό των ε, μέσων που βρίσκονται στην τροχιά είναι η μόνη, ε, το μόνο μέσο που βασίζεται σε συνθήκη για να αναπτύξουμε, να έχουμε μια πλήρη παρατήρηση του διαστημικού χώρου. Εμείς διαχέουμε τις πληροφορίες σχετικά με την ανάκτηση ε, σωμάτων από το διάστημα, δορυφορικών σωμάτων που χρησιμοποιούν πυρηνική ενέργεια, ε, περί τα 9.000 ε, σώματα έχουμε καταγράψει από το 2007, άνω του 20% των οποίων στα τελευταία 6 χρόνια έχουν τεθεί στη ροχιά. Έχουμε δηλαδή, αν θέλετε, μια εχμή στην, ε, στο γράφημα, στην καμπύλη αυτή τη στιγμή. Οι κατευθυντήριες γραμμές πάντως είναι μια, ένα πολύ καλό παράδειγμα του πώς το διάστημα μας εξωθεί σε ένα σύστημα πολυμέρειας και της πολύ μεγάλης παράδοσης που έχουν τα Ηνωμένα Έθνη για την ειρηνευτική χρήση ε, του διαστήματος όπως κάθε άλλου χώρου σε ειρηνικά πλαίσια. Έχουμε όμως πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε. Ε, πρέπει να έχουμε περισσότερες ε, προσπάθειες για να εφαρμόσουμε το παρόν ρυθμιστικό και νομικό πλαίσιο. Παρέχουμε συμβουλές σε κρατικούς και μη κρατικούς φορείς σχετικά με την ικανότητα εκτόξευσης που μπορούν να έχουν, σχετικά με την νομική τους ε, ε, γνώση και πλαισίωση και υιοθετώντα αυτή την προσέγγιση, την προσέγγιση bottom-up προσπαθούμε να εντοπίσουμε τις χώρες που χρειάζονται περισσότερο τη βοήθειά μας. Η πρώτη χώρα και η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που συνεργάστηκε με την UNOSA ε, ήταν το Λουξεμβούργο για την ανάπτυξη ε, τεχνολογικής ε, και άλλης βοήθειας που μπορεί να παραχθεί στις χώρες. Συμπερασματικά θέλω να πω ότι στα Ηνωμένα Έθνη ε, διατηρούμε ένα, μια οπτική παγκόσμιας εμβέλειας μια συνεργασία ολιστική με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα, θα ήταν πολύτιμη βοήθεια για μας. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Θα περάσουμε τώρα στη συζήτηση και θα δώσω το λόγο σε όσους τον ζήτησαν και σας παρακαλώ να είστε σύντομοι. Έχουμε ξεπεράσει λίγο την ώρα, οπότε μάλλον θα πάμε μέχρι τις 10.45 αντί για 10.30 για να απαντηθούν και οι ερωτήσεις σας. Θα κάνουμε ένα πρώτο γύρο ερωτήσεων και οι ομιλητές μας θα απαντήσουν ό,τι επιθυμούν στις ερωτήσεις που επιθυμούν να απαντήσουν για να αποφύγουμε επαναλήψεις που καμιά φορά γίνεται βαρετές αν απαντούν όλες σε όλες οι ερωτήσεις. Ο κύριος Οστρεβίσιος της ομάδας Renew Europe πρώτος. Thank you, Chair. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και όλους τους προσκεκλημένους για τις ε, πολύ ενδιαφέρουσες και λεπτομερείς παρουσιάσεις. Έχω τα εξή ερωτήματα. Καταρχά, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προσπαθούμε να θεμελιώσουμε το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα σε θέματα πολιτικής ε, του διαστήματος. Αλλά υπάρχει ένα κενό προς το παρόν ε, στον ε, συντονισμό. Υπάρχει έλλειψη δηλαδή επενδύσεων έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε καλύτερα αποτελέσματα για το μέλλον. Έπειτα, η διαστημική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποιο βαθμό διασυνδέεται με την ε, αμυντική τεχνολογία. Είμαστε υπό Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας και οφείλουμε να δούμε αυτήν την ε, σχέση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να υιοθετήσει και αυτή τη διάσταση και να τη χρησιμοποιήσει στην ε, διαστημική της και αμυντική της πολιτική, να χρησιμοποιήσει δηλαδή τις σχετικές τεχνολογίες. Τρίτον, Γνωρίζουμε ότι είμαστε μεν καλοί, αλλά όχι καλύτεροι σε όλα. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω σε ποιο βαθμό εξαρτώμαστε από τις χώρες εταίρους και τη δική τους συνεισφορά στην διαστημική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμείς οι ίδιοι. Τι είδους συνεργασία έχουμε με εταίρους όπως το Ισραήλ και η Ουκρανία χώρες οι οποίες έχουν ε, ικανότητες τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Και τέλος, ε, μια που είμαστε και στην ε, Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας, να πω ότι πρόσφατα άκουσα για τις διαστημικές τεχνολογίες αναγνώρισης ως κάτι το καλό. Γνωρίζουμε όλοι το σύστημα Galileo, όμως τι γίνεται με τις ε, παράνομες προσεδαφίσεις ε, ρωσικών σκαφών στα νησιά της Νορβηγίας ε, που αναφέρουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Το σύστημα που χρησιμοποιούν εντόπισε αυτές τις παράνομες προσεδαφίσεις σε έδαφος Νορβηγίας. Εμείς είμαστε ικανοί να κάνουμε κάτι αντίστοιχο ή όχι. Ευχαριστούμε. Δίνουμε τώρα το λόγο για το ΕΛΚ στον Μιχαήλ Γκάλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω γερμανικά. Παρατηρώντας λοιπόν όλα αυτά που έχουμε στην ημερήσια διάταξη και έχοντας ακούσει τις τέσσερις πολύ εντυπωσιακέ παρουσιάσεις των προσκεκλημένων, βλέπω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τοποθετηθεί, έχει τοποθετηθεί εδώ και χρόνια για αυτά τα θέματα. Νομίζω πως ε, πρέπει πραγματικά να αναλάβουμε από κοινού δράση, διότι είναι πολύ επίπεδο το θέμα, έχει πολλές ε, διαστάσεις και νομίζω πως δεν χώρα ε, περιθώριο για εθνικές τακτικές. Χρειάζεται από κοινού να δούμε πώς ε, θα δράσουμε, τι επιλογές έχουμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι στον ε, τομέα αυτό οφείλουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό. Και ιδιαίτερα, μια που αναφέρθηκε το Γκαλιλαίο, να δούμε τι γίνεται με τον ε, προϋπολογισμό. Όταν εξετάζουμε θέματα συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, υπάρχουν ορισμένα, ορισμένες λεπτομέρειες που πρέπει να εξετάσουμε. Βέβαια, πρέπει να φροντίσουμε να ε, πρόκειται για πολιτικό χαρακτήρα των εφαρμογών και όχι στρατιωτική ε, χρήση αυτών των τεχνολογιών. Δεν ξέρω λοιπόν αν θα άξιζε τον κόπο να εξετάσουμε και στρατιωτικές εφαρμογές ε, των ε, τεχνολογιών διαστήματος. Οι καιροί αλλάζουν, όπως ακούσαμε και από την κυρία Κλάις. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να τη ρωτήσω αν θα μπορούσε να μας πει με περισσότερες ε, λεπτομέρειες τι προβλέπεται από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Πέραν αυτών, η άλλη ερώτηση που έχω να κάνω αφορά κυρίως ευρωπαϊκό περιεχόμενο, δηλαδή σε... Ε, δηλαδή πού βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση, αν υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα, κάποιο ταμείο, το ε, άμυνα στο οποίο προβλέπεται να συσταθεί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε όλα αυτά που λέμε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε στο έπακρο όλες τις ε, δυνατότητες που διαθέτουμε, διότι οι δυνατότητες υπάρχουν, πολιτική βούληση όμως μας ε, λείπει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για το ID η κυρία Μπομφρίσκου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω Ιταλικά. Να εκφράσω την εκτίμησή μου για την ποιότητα και τον πλούτο των παρουσιάσεων που ακούσαμε. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση για μια διευκρίνηση στους ομιλητές όσον αφορά την εμπειρία του Γαλιλαίου και του Κοπέρνικου που αναφέρθηκαν τόσο πολύ σε θέματα προστασίας των δικών μας ε, διαστημικών στοιχείων. Πώς μπορούμε να εξάγουμε την εμπειρία από το Κοπέρνικου και τον Γαλιλαίο σε άλλα διαστημικά προγράμματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση Και τα διαστημικά προγράμματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω. Ε, μόλις υπενθύμησε ο συνάδελφος Γκάλερ έχουν πολιτικό χαρακτήρα ή είναι απλά αποτέλεσμα της ανάπτυξης ε, των τεχνολογιών και της τεχνογνωσίας. Ευχαριστώ. Merci. Ευχαριστούμε κύριε Κρούντλερ για το Ρηνιού. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μια μικρή σκέψη σήμερα το πρωί για το διαστημικό δόγμα. Η κυρία Κλάς μίλησε για τη συνθήκη για το διαστημά του 1967 που απαγορεύει τη χρήση πυρηνικών όπλων στο διάστημα, ε, όπλα μαζικής καταστροφής ε, στο διάστημα, σε ε, τροχιά στο φεγγάρι, αλλά δεν απαγορεύει τα κλασικά μέσα. Σήμερα το διάστημα ε, και η επιτήρηση έχουν διάφορες δυσκολίε, ε, Υπάρχει στρατιωτικοποίηση αναγνωρισμένη πλέον κάπου και όλο και περισσότερο υπάρχουν κίνδυνοι στρατιωτικοποίηση του διαστηματο Κατά την άποψή σα. η απόφαση του Πρόεδρου Τραμπ, όπω ανακοινώθηκε τον Ιούνιο του 2018, να δημιουργήσει το Space Force του, τη διαστημική του δύναμη, όχι μόνο για να δίκει το διάστημα, αλλά είναι μια πραγματική στρατιωτική δύναμη. Ε, ναι, δύναμη είναι αλλαγή του ε, διαστημικού δόγματος ε, πέραν τη επιτήρησης και η Ευρώπη μπορεί να αναλάβει κάποια πρωτοβουλία για να εμποδίσει αυτή την πρωτοβουλία, τη στρατιωτικοποίηση. Η άποψή μου ε, στο πλαίσιο του διαστημικού κανονισμού τα 16,9 δις ευρώ που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να επικυρωθούν στο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο για να έχουμε τα μέσα να μαχηθούμε, για να το πω έτσι, στο διάστημα για να επιβάλλουμε πιο ειρηνικέ λύσει. Υπάρχει ανάγκη να είναι παρόν αυτό ο προπολογισμό για να δράσει αποτελεσματικά η Ευρώπη. Ευχαριστούμε. Και τέλο για το ΕΛΚ, ο κ. Πέτερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους προσκεκλημένους, διότι ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε. Έχω μία ερώτηση για τη σχέση μεταξύ Ηνωμένων Εθνών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω πως ήδη ε, ακούστηκε ότι η πολυμέρεια είναι πάρα πολύ σημαντική για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό στο μέλλον, όμως γνωρίζουμε ότι αυτή η ιδέα δεν έχει και τόσο μεγάλη επιτυχία, ότι υπάρχουν μεγάλοι παίκτες όπως η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες που δεν είναι Γι' αυτό η ερώτησή μου είναι πώς μπορούμε στο μέλλον να εξασφαλίσουμε ότι οι συζητήσεις εντός των ε, Ηνωμένων Εθνών θα έχουν βαρύτητα. Εδώ να ευχαριστήσω το, εσάς και το έργο σας, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την διατήρηση αυτής της πολυμέρειας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Δίνω λοιπόν το λόγο στους ομιλητές μας. Θα πρότεινα ο καθένας να πάρει το λόγο για τρία με τέσσερα λεπτά το πολύ. Ξεκινάμε από εσάς κύριε Ζαϊκ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Ας αφήσουμε στο πλάι τα τεχνικά ζητήματα. Οι συναδελφοί μου είναι σε καλύτερη θέση από μένα για να απαντήσουν. Ήθελα να πω δύο λόγια για το ζήτημα της, ε, του πολυμερού συστήματος σε σχέση με το διάστημα. Όπως μας δείχνει η ιστορία, η υλοποίηση πλαισίων ισορροπίας και ελέγχου ε, βάσει πολυμερούς προσέγγισης ανέκαθεν γίνονταν από αξιόπιστους και σεβαστούς φορείς σε θέματα άμυνας. Ε, η πολυμερής προσέγγιση, το πλαίσιο ε, το, στο οποίο είχαμε ε, μια ασφαλή προσέγγιση για πολλά χρόνια και που σήμερα ε, δέχεται επίθεση, αμφισβητείται ή ε, καταστρέφεται, είχε δημιουργηθεί ιστορικά από φορεί αξιόπιστους, δυνατούς στον τομέα της άμυνας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλει να επανοικοδομήσει πολυμερές σύστημα το οποίο θα λειτουργεί για ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα, αυτό θα είναι δυνατόν μόνο, θα λειτουργεί στον τομέα τη αμυνα η ευρωπαικη ενωση αν θελει να επανοικοδομησει πολυμερε συστημα το οποιο θα λειτουργει για ολοκληρη τη διεθνη κοινοτητα αυτο θα ειναι δυνατον μονο πιστευω αν δειξει αξιοπιστια στον τομεα τη αμυνα Ο διαστημικό τομέα και κλείνω εδώ, είναι, δεν είναι παρά μια ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για το μέλλον, για τις μελλοντικέ γενιές. Είναι μια ευκαιρία να οικοδομήσει μια αξιοπιστία στρατιωτικές δυνατότητες που θα εξυπηρετήσουν την ειρήνη ε, και τις πολυμερείς μας ισορροπίες έτσι ώστε να ηγηθούμε στον τομέα αυτών. Δεν μπορούμε να υπολογίζουμε στι δυνατότητε άλλων και να βασιζόμαστε σε αυτέ, ούτε να αναθέτουμε σε τρίτου τι δυνατότητέ μα, ακόμη και αν είναι σύμμαχοι ή στον ιδιωτικό τομέα. Δεν μπορούμε να αναθέτουμε στον ιδιωτικό τομέα ε, τέτοιε δυνατότητε για να χτίσουμε την πολυμερή προσέγγιση. Το διάστημα λοιπόν από αυτή την άποψη, για να απαντήσω στην τελευταία σα ερώτηση, είναι μια τεράστια ευκαιρία ε, που θα επιτρέψει στην Ευρώπη να ε, επιβεβαιώσει τον πολιτικό τη εθελοντισμό. Πάντα μιλάμε για τη SpaceX και τη New Space. Σήμερα το εισιτήριο για τον πυραυλό Falcon 9 είναι 99 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ ανταγωνιστικό. Μην ξεχνάμε ότι το Falcon 6 υπάρχει διότι η ΕΠΑ, το Αμερικανικό κράτος, επιχορήγησε το Falcon 6 με 360 εκατομμύρια ευρώ. Αν δώσουμε λοιπόν τις ίδιες δυνατότητες στους δικούς μας φορείς, ε, υπάρχει τέτοια πολιτική στήριξη γιατί υπάρχει η βούληση και η ενσυνείδηση. Για να μπορέσουμε να υπερασπίσουμε αύριο λοιπόν την πολυμερή προσέγγιση ως Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πρέπει να ξεχνάμε και αυτή την πραγματικότητα. Ευχαριστούμε. Δίνω το λόγο στην κυρία Καρίν Κλέση γιατί ξέρω ότι έχετε πολύ φορτωμένο πρόγραμμα σήμερα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε τα τεχνικά ερωτήματα θα τα αφήσω στον συνάδελφο της GSA. Ε, πράγματι θεωρώ ότι η απόφαση του Προέδρου Τραμπ να αναπτύξει μια διαστημική δύναμη αλλάζει τελείως τα πράγματα, την ισορροπία αλλά και η πιθανή απόφαση του ΝΑΤΟ να καταστήσει το διάστημα νέο πεδίο στρατιωτικού ανταγωνισμού επίσης αλλάζει τελείως το παιχνίδι. Γιατί πρόκειται για ένα νέο πολεμικό πεδίο δυνητικά το οποίο θα άλλαζε τα πάντα. Ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς το παρόν μην υπάρχει μια ομοιομορφία απόψεων μεταξύ των κρατών μελών για το τι πρέπει Πώ πρέπει να διαμορφωθεί το μέλλον σε αυτά τα θέματα. Έχουμε δει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού τη γαλλική και την ιταλική κυβέρνηση να έχουν προχωρήσει σε σημαντικές δηλώσεις σχετικά με την αμυντική τους δυνατότητα και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό ως πρώτο βήμα. Τώρα βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζεται και εξαρτάται στρατιωτικά και αμυντικά από τα κράτη-μέλη και η πολιτική θέση των κρατών μελών από αυτού δεν είναι καθόλου ομοιόμορφη προς το παρόν. Επομένως έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας και υπάρχουν κάποιοι άξονες δραστηριότητες που έχουν αναλυφθεί στα πλαίσια των ΠΕΣΚΟ, της ε, συνεργασίας ε, στην, ε, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας για την ανάπτυξη κάποιων δυνατοτήτων, κάποιου δυναμικού, το οποίο δείχνει μία οδό προς τα εμπρός, αλλά θα πρέπει να έχουμε μια μεγαλύτερη ομοιομορφία απόψεων προκειμένου πραγματικά να ξεκινήσουμε κάτι αυτό. Για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και συστήματος πολυμερίας ε, ε, είναι και αυτό μέρος του γενετικού κώδικα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πεδίο που η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και πρέπει να είναι πολύ ενεργή μαζί με τα κράτη της μέλη και στα πλαίσια του κόπουος θα μπορούσαν να υιοθετηθούν οι 21 κατευθυντήριες γραμμές που είχαν υιοθετηθεί τον Ιούνιο όπου οι ευρωπαϊκοί φορείς μπορούν να, να καταδείξουν με την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών ότι είναι μέρος του συστήματος πολυμέρειας να δείξουν δηλαδή με απτό τρόπο, να δώσουν ένα παράδειγμα, το οποίο θα ενίσχυε την διαφάνεια και την ανάπτυξη εμπιστοσύνης. Θα ήταν ένα σαφές βήμα δηλαδή προς μια ανάκτηση, αν θέλετε, των στήματων πολυμέρειας διεθνώς. Θα έμενα εδώ και ίσως ε, θα έδινα στον συνάδελφο της ε, GSA το λόγο για τα πιο τεχνικά. Ο κύριος Κλοντέλ, ευχαριστώ πρόεδρε. Σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας και τεχνολογίας, σε σχέση με τον κύριο Ζαζόεκ, ε, να πω τους δύο βασικούς ανταγωνιστές που είναι η ΙΠΑ, ε, όπου βλέπουμε ότι ε, αναγκαζόμαστε να είμαστε πολύ πιο καινοτόμοι με τη στάση που τηρούν οι Ηνωμένε Πολιτείε με τα μέσα συλλογής πληροφοριών, παρατήρησης και τα λοιπά, έρευνας, αλλά χρειάζεται και ένα ελάχιστο υποστήριξη της ε, βιομηχανίας μας, ώστε να μείνει ανταγωνιστική, να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε ανταγωνιστικά προϊόντα για την ε, προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το παράδειγμα του ΣΠΕΞΙΣ ε, που μόλις αναφέρθηκε ε, υπάρχουν και του SpaceX μάλλον ε, που είναι υπό το Υπουργείο Αμήνης των πολιτειών με συγκεκριμένες παρα... εντολές παραγγελίας, πλαίσια παραγγελιών με πολύ υψηλές τιμές, ε, με μέσα πολύ υψηλή ταχύτητα ε, του διαδικτύου για παράδειγμα, δορυφορικά μέσα. Οι Αμερικανοί πρότειναν ε, τον εξοπλισμό πολιτικών δορυφόρων με στρατιωτικά συστήματα. Δηλαδή βλέπουμε ότι δεν έχουμε ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού με τους Αμερικανούς ως προς αυτή τη στάση. Δεν τηρούμε την ίδια στάση. τα κράτη-μέλη ε, ελέγχουν, θα έλεγα, και τα θεσμικά όργανα. Πρέπει να έχουμε λοιπόν ένα κοινό πολιτικό προσανατολισμό και συντονισμένο για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Στο επίπεδο του Κοπέρνικους, ναι, μπορούμε να εφαρμόσουμε ε, τη γνώση που έχουμε συλλέξει μέσω του Γκαλιλαίου για τη διάχυση των δεδομένων για τις γνώσεις, η οποία προς το παρόν είναι ελεύθερη και δωρεάν. Επομένως μιλούμε για ένα κρυπτογραφημένο σύστημα από τη μία μεριά και ένα open system από την άλλη. Τώρα, με την γνώση που έχουμε ανακτήσει επί του Γκαλιλαίου θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε και εμείς σε ένα ανοιχτό και ένα κλειστό σύστημα δεδομένων. με κλίδα που θα μπορούσαμε να δώσουμε στα κράτη-μέλη ώστε να μην έχουν πρόσβαση οι ανταγωνιστές μας σε ευαίσθητα δεδομένα. Υπάρχει και αυτή η διπολικότητα που αναφέρθηκε, δεν έχουμε τον ίδιο προεπολογισμό. Η βιομηχανία βασίζεται στην πολιτική δραστηριότητα και έχουμε υποβαθμίσει την διακυβερνητική συνεργασία, την αμυντική στο πεδίο αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Για να κλείσουμε η κυρία Διπίπου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ εν συντομία στην πολυμερή προσέγγιση και το ρόλο των Εθνών και πιθανές συνεργίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρθηκε ήδη αυτό το ισχυρό αποτέλεσμα της Επιτροπής για την Ελληνική Χρήση του διαστήματος. Ε, ε, τον Ιούνιο φέτος, μετά από κάποια χρόνια δουλειά, ανέκριναν το προημείο και τις πρώτες 21 κατευθύντηρες γραμμές για την ε, μακροχρόνια βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων στο απότερο διάστημα. Η διαδικασία είναι τέτοια που οι αποφάσεις λαμβάνονται με συνένεση, δηλαδή χωρίς ψηφοφορία. Αυτό σημαίνει ότι οι κατευθυντήρες γραμμές έχουν συζητηθεί από όλα τα μέλη της Επιτροπής ε, κατά λέξη για ένα χρονικό διάστημα. Όλοι λοιπόν έχουν δεσμευτεί ε, να τη στηρούν. Κάποιες κατευθύντηρες γραμμές ε, δεν οδήγησαν σε επίτευξη συνένεσης και τώρα έχουμε μια νέα ομάδα εργασίας για την υλοποίηση αλλά και για τη συζήτηση του πώς θα συνεχιστεί τι θα γίνει στη συνέχεια όσον αφορά τη διαδικασία έγκρισης για επιπλέον κατευθύντηρες γραμμές. Δεν είναι λοιπόν ε, υποχρεωτικές, δεν είναι δεσμευτικές, αλλά ταυτόχρονα είναι αυτό που θέλουν να κάνουν τα κράτη-μέλη. Κάτι σημαντικό είναι ότι στην Επιτροπή Ειρηνικών Χρήσεων του Απότρου πριν πέντε χρόνια, όταν εγώ ανέλαβα διευθύντρια στο γραφείο μου, είχαμε 76 μέλη σε πέντε χρόνια από 76 πήγαμε στα 95 μέλη. Ε, αρκετά μεγάλη αύξηση που σημαίνει ότι αυτή η Επιτροπή για τις Ειρηνικές Χρήσεις ε, του Εξώτερου Διαστήματος είναι η πιο ταχύως αναπτυσσόμενη Επιτροπή. Και δείχνει επίσης ότι το διάστημα αποκτά όλο και μεγαλύτερη σπουδαιότητα για πολλές χώρες. Καλύπτουμε με 95 μέλη, λίγο πάνω από 6 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Οι χώρες... Έχουμε και μια περιοχή που δεν εκπροσωπείται επαρκώς και είναι η Αφρική. Στην Κόπους ε, συνεργαζόμαστε λοιπόν στενά με τα σημερινά κράτη-μέλη για να μπορέσουμε να φέρουμε όλο και περισσότερες χώρες ε, στο τραπέζι της συζήτησης. Γιατί, διότι πρώτα απ' όλα είναι σημαντικό να έχουμε μια συνείδηση, ευαισθητοποίηση, να παρέχεται διαφάνεια, όλα τα κράτη-μέλη να μπορούν να κατανοήσουν τι συμβαίνει στις άλλες χώρες. Και δεύτερον, θέλουμε να έχουμε υπόψη μας, και αυτό είναι σημαντικό πιστεύω παντού, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο εμπορικός κλάδος προχώρα με τεράστια άλματα και τα θεσμικά όργανα ε, δεν μπορούν απαραίτητα να ακολουθήσουν με την ίδια ταχύτητα. Κάποιοι τομείς, η διαχείριση της διαστημικής κίνησης ή η, ο εντοπισμός θέσης στο διάστημα και σε αυτούς ε, τους τομείς ε, οι ταχύτητες, οι, οι δραστηριότητες, οι εμπορικές γίνονται με μεγάλη ταχύτητα, οπότε... Το να διασφαλίσουμε κάποιο διαστημικό χώρο είναι σημαντικό για να μπορέσουν να διατηρήσουν την ειρηνική χρήση του διαστήματος στα κράτη με μια πολυμερή προσέγγιση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχω παρά να ευχαριστήσω τους ομιλητές για την ποιότητα των παρουσιάσεών τους. Ε, παρατηρούμε ότι τα μέλη της Υποεπιτροπής ε, έχουν σαφέστατα μεγάλο ενδιαφέρον. Ε, θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν για την παρουσία σας. Πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε τέτοιες ακροάσεις για να εξετάσουμε τις ευκαιρίες που μας δίνει το διάστημα και η διάσταση άμυνας και ασφάλειας στο διάστημα. Ξανά ευχαριστώ και πάλι τους ομιλητές. Συνάδελφοι, να επανέλθουμε στις εργασίες του πρωινού με την ανταλλαγή επόψεων που έχουμε για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Παρέμβασης. Όσοι επιθυμούν να συζητήσουν, παρακαλώ να το κάνουν εκτός της αιθούσης και θα ήθελα να καλασορίσω τον στρατηγό Μπρίνο Φουσάρ, επικεφαλής ε, του ευρωατλαντικού κλάδου του επιτελείου γαλλικού στρατού, τον ε, στρατηγό Ματ Πίρσον, εκπρόσωπο του ΝΑΤΟ, και τον ε, συνταγματάρχη Άιν Ρέκαντ, ε, επιτετραμένο του Εστονικού Υπουργείου Αμήνης. Είχαμε από το 2018 την υπογραφή μια επιστολής ε, προθέσεων από τη Γερμανία, το Βέλγιο, τη Δανία, την ε, Γαλλία, την Εστονία, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, αν ακούσαμε όλες τις δηλώσει καλά. Η Ιταλία επίσης, όπως και η Ελλάδα, εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την ανάδειξη ενός κοινού πλαισίου μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών που συμμερίζονται την πολιτική βούληση και τις αμυντικές στρατιωτικές δυνατότητες για επιχειρησιακή δέσμευση. Το 2019 η πρωτοβουλία ε, πέρασε μια φάση ανάπτυξης ε, με ένα πρώτο κύκλο εργασίας. Ε, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε σχετικά με τις δραστηριότητες που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα και να μα ενημερώσετε επίσης για τις επόμενες φάσεις. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Παρέμβασης είναι ένα νέο πλαίσιο καινοτόμο και συμπληρωματικό και τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΝΑΤΟ. Θα θέλαμε λοιπόν το όραμα το δικό σα για τις συνέργειες μεταξύ της πρωτοβουλίας και των διαφόρων άλλων πλαίσιων συνεργασία κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον στρατηγό Φουσά για ένα δεκάλεπτο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε μεγάλη μου τιμή σήμερα να σας μιλώ για ένα θέμα πολύ σημαντικό που είναι πολύ σημαντικό για τον πρόεδρο Μακχόν και που μας αφορά όλους ε, και εμάς και τις μελλοντικέ γενιές. Τώρα, γιατί η πρωτοβουλία παρέμβασης. Είναι μια πρωτοβουλία υπό τον πρόεδρο Μακχόν στην ομιλία στη Σορβόνη ε, το 2017 για μια ισχυρή πολιτική βούληση ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Άμυνας με τριπλή παρατήρηση συμπέρασμα ότι οι κρίσεις στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Υπήρου αφορούν άμεσα στην ασφάλεια των πολιτών και πολλαπλασιάζονται, γίνονται οξύτερες και πιο περίπλοκες. Δεύτερη παρατήρηση, έχουμε διάφορες, πολλές και διάφορες προκλήσεις και προβλήματα αλλά και πολλά μέσα στη θέση μας που δεν χρησιμοποιούμε. Και επομένως έχουμε μια δυσκολία συνεργασίας σε νέα θέατρα επιχειρήσεων. Ε, αναφέρω απλώς ε, το Μαλή ε, ως παράδειγμα. Έχουμε ανάγκη ανάπτυξης της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι είμαστε υπερβολικά εξαρτημένοι από συμμάχους όπως οι Αμερικανοί. Αυτό είναι το πλαίσιο εντός του οποίου λοιπόν η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Παρέμβασης εκκίνησε με απότερο στόχο να διαφωλύνει και να επιταχύνει την ανάληψη δεσμεύσεων προλαμβάνοντας μελλοντικές κρίσεις και ο βασικός μοχλός της πρωτοβουλίας είναι να πολλαπλασιάσει την κοινή στρατηγική προσπάθεια των χωρών που έχουν τη δυνατότητα αυτή και που έχουν και τη βούληση ανάπτυξης στρατιωτικών δυνάμεων σε εξωτερικές παρεμβάσεις. Μιλούμε για μια προοδευτική αυξανόμενη συνεργασία εφόσον θα έχουμε εγκαθιδρύσει αυτή την κοινή βούληση συνεργασίας στρατιωτικής και αμυντικής. Ε, αυτά είναι μέτρα που θα αύξαναν την εμπιστοσύνη ε, μεταξύ των κρατών μελών ώστε να αναλυθεί ενδεχομένως μια κοινή στρατιωτική δυνατότητα και βούληση της ανάληψής της. Από την εκκίνηση της πρωτοβουλίας όλοι οι εταίροι, όλοι οι συνεργάτες και είμαι σίγουρος ότι οι συνάδελφοι στα αριστερά μου θα το βεβαιώσουν ε, μιλούν για την ευελιξία της, για την ρεαλιστική της προσέγγιση της και για το επίπεδο της εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται μεταξύ των κρατών μελών. Κάτι που αυξάνεται έντονα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εννέα ήταν τα αρχικά μέλη της πρωτοβουλίας τον Ιούνιο του 2018 Γαλλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ε, Γερμανία, Ολλανδία, Εστονία και Δανία. Και περάσαμε στους 10 με την ε, έλευση της Φινλανδίας και τελικώς 12 μετά την υπουργική του Σεπτεμβρίου ε, του περασμένου Σεπτεμβρίου και ίσως να είμαστε και στους 13 μετά τη Σουηδία λοιπόν ίσως και η Ιταλία να συμμετέχει και Άλλε χώρε έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, έντονο ενδιαφέρον για την πρωτοβουλία αυτή, για τη συνεργασία αυτή. Τώρα, πρωτού αναφερθώ στις εργασίε ε, που, που έχουμε υλοποιήσει μέχρι σήμερα, θα σα αναφέρω αυτό που αναφέρουμε battle rhythm της πρωτοβουλίας, το ρυθμό δραστηριότητά τη και το ρεαλισμό της προσέγγιση αυτή. Έχουμε συνήθως μια συνάντηση στην αρχή του κύκλου, συνήθως Σεπτέμβριο, ή Οκτώβριο, μετά δύο συναντήσεις των επιτελεαρχών ή των εκπροσώπων των επιτελείων, που είναι οι συζητήσεις των στρατατικών επιτετραμένων και μετά ένα πολιτικό κύκλο συζήτησης ε, για την προετοιμασία, για την προετοιμασία με της επόμενης της ακόλουθης υπουργικής. Έχουμε επίσης ομάδες εργασίας θεματικής ή γεωγραφικής εξέτασης για τις στρατιωτικές θεματικές, κάθε κράτος μέλος μπορεί να προτείνει νέα θεματική ή νέα ομάδα εργασίας. Η μόνη δέσμευση για τη δημιουργία μιας ομάδας εργασίας είναι ότι πρέπει από την αρχή να καταδεικνύει ότι δεν θα έχει επικαλύψεις με ε, τον ΝΑΤΟ, ε, τον ΟΑΣΑ ή οποιονδήποτε άλλο διεθνή οργανισμό ή πλαίσιο. Έχουμε τέσσερις βασικές γραμμές οριζόντιας συνεργασίας στρατηγική συνεργασία και ανταλλαγή δεδομένων, ε, ανάπτυξη σεναρίων, υποστήριξη επιχειρήσεων και ε, συλλογή εμπειρίας. Έχουμε οκτώ σήμερα ομάδες εργασίας, ε, τέσσερις γεωγραφικής, για το Σαχέλ, την Καραϊβική, την Βαλτική και τον Ινδικό ωκεανό. Τέσσερις θεματικές ομάδες εργασίας για την, ε, για τα επίπεδα ισχύω, την τρομοκρατία, την εξωτερική επιρροή στην Αφρική και νομικές υποθέσεις. Αυτές συνέρχονται όσο τακτικά χρειάζονται υπό την επικουρικότητα, χωρίς λεπτομέρειες ε, θα σας περιγράψω λίγο τις ομάδες αυτές. Για το Σαχέλ. Εδώ η πρόθεση είναι ο συντονισμός και η συνεργασία στα θέματα που αφορούν στην περιοχή αυτή, είτε για εθνικές επιχειρήσεις όπως οι γαλλικές, είτε επιχειρήσεις όπως εκείνη του Μαλή ή ε, συνοριακών περιοχών συνεργασίας. Για την ε, ομάδα της Καραϊβικής είχαμε ας πούμε τον τυφώνα Ήρμα, την συνεργασία και το συντονισμό στην αντιμετώπιση δηλαδή καταστροφών φυσικών. Χαρτογράφηση των ε, φορέων των επιχειρησιακών που έχουμε νομικού πλαισίου, του περιφερειακού επίση για να έχουμε πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση σε μελλοντικέ κρίσει. Στην ομάδα Βαλτική, μιλούμε για τα διακυβεύματα τη περιοχή σε επίπεδο διπλωματικό και τακτικό για να συντονίσουμε την ανταπόκρισή μας στο μέλλον. Για τον Ειδικό Ωκεανό μιλούμε για τη φιλοδοξία της ε, ε, δημιουργία μια καλύτερη χαρτογράφηση τη κατάσταση στην περιοχή, τα σενάρια κρίσεων, επί τη βάση των πληροφοριών που έχουμε για τους αναδυόμενους φορείς και ο συντονισμός των στρατιωτικών επιτελείων για να αντιμετωπίσουν αυτά. Για το επίπεδο των δυνάμεων. Εδώ μιλούμε για αμοιβαία υποστήριξη σε περίπτωση ε, στρατιωτικής επιχείρησης εκτός Ευρώπης, ιδιαίτερα υπό τις επιχειρήσεις Χάμιλτον και Σαντεάν στη Συρία ε, και άλλες εφόσον χρειαστεί. Ε, ε, στην ομάδα αντιτρομοκρατίας έχουμε ένα ετήσιο σεμινάριο. Το επόμενο θα είναι 15 Νοεμβρίου στο Παρίσι. Ε, η ομάδα Αφρικής εστιάζεται στους μη ευρωπαϊκούς φορείς και τη δεθεότητα στην Ήπειρο αυτή για τα στρατιωτικά επίπεδα δύναμη στην Αφρική. Η νομική ομάδα συνέρχεται ανάλογα με την ανάδειξη του κάθε θέματος ενδιαφέροντος και όπως εξελίσσεται το διεθνές νομικό πλαίσιο. Προσπαθούμε λοιπόν να εστιαστούμε σε ανθρωπιστικές επιχειρήσεις ή σε ζώνες ιδιαίτερο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που σήμερα δεν καλύπτουμε ή που καλύπτουμε μόνο μερικώς. Δύο σημαντικά ζητήματα συνολικά είναι τα εξή. Πώς εξελίσσεται η σε ζωνες ιδιαιτερο ευρωπαικου ενδιαφεροντος που σημερα δεν καλυπτουμε η που καλυπτουμε μονο μερικω δυο σημαντικα ζητηματα συνολικα ειναι τα εξη πως εξελισσεται η πρωτοβουλια η ποιοι θα είναι οι νέοι εταίροι ενδεχομένω, πώς τη φανταζόμαστε σε κάποια χρόνια στο μέλλον. Για την πιθανή της προέκταση δεν είναι ο στόχος μας η διεύρυνση χωρίς να είμαστε όριμοι γι' αυτό. Έχουμε, ένα κριτήρια, έχουμε κριτήρια εισόδου αρκετά αυστηρά, τουλάχιστον να είναι κανείς μέλος δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΝΑΤΟ, προτού να έχει επιχειρησιακές δυνατότητες δηλαδή, ε, εκτός των συνόρων. Όλα αυτά γίνονται συνδετικά και υπό του υπουργού αμήνη των χωρών τη πρωτοβουλία για το μέλλον. Ρεαλιστικά, αν είναι να δώσουμε μια εκτίμηση των ε, μελλοντικών κρίσεων, η πρωτοβουλία θα έπρεπε στο πιο φιλόδοξο σενάριο, σε περίπτωση ανάγκης να επιτρέψει στρατιωτική ανάπτυξη εκτός ευρωαϊκών συνόρων, με τα μέσα που θα επιτρέπουν οι χώρες που θα έχουν συνενέσει με την πολιτική συνένεση, με την πολιτική βούληση των ηγεσιών τους και έχοντας συνεργαστεί με, τις, ε, με τους πολυμερείς ε, φορείς ώστε να έχουμε όλα τα μέσα στη διάθεσή μας για να αποφασίσουμε αν ναι ή όχι πρέπει κάπου να παρέμβουμε στρατιωτικά και τι δυνάμεις θα χρειάζονταν, τι επιχείρηση θα ήταν, ποιοι θα συμμετείχαν κτλ. Τώρα για τις αντιμετωπίσεις ε, κρίσεων η πρωτοβουλία ε, θα μπορούσε να επιτρέψει καλύτερη υποστήριξη, αμοιβαία βοήθεια για ε, υπηκόους ε, ευρωπαϊκών χωρών που βρίσκονται σε κάποια μακρινή χώρα, για παράδειγμα, ε, ή σε περίπτωση απειλής και πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Η κινητοποίηση στα πλαίσια της πρωτοβουλίας παρέμβασης είναι νομίζω μια συλλογική συνείδηση ότι δεν μπορούμε να δρούμε μόνοι μας, δεν μπορούμε να δρούμε κατακαιρματισμένα, αντιμετωπίζουμε απειλές που δεν ε, κάνουν διακρίσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η σχέση μας ε, με τον στρατηγικό σύμμαχο των Πολιτειών, ε, η κατάσταση των σχέσεών μας και η μελλοντική της τάση καθιστά απαραίτητο να συνεργαστούμε. Είμαι απολύτως διάθεσή σας να απαντήσω σε ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ στρατηγή. Δίνω τώρα το λόγο στον ε, ταξιέρχο Ματ Πίρσον. Σας ευχαριστώ πολύ. Με μεγάλη μου χαρά βρίσκομαι σήμερα ενώπιόν σας για να σας μιλήσω λοιπόν για το θέμα μας. Θα ήθελα να πω καταρχάς όσο προς την πορεία του Ηνωμένου Βασιλείου ότι βρισκόμαστε σε διαδικασία εκλογών και αυτά που μπορώ να σας πω είναι κάποιες σκέψεις και κάποιοι προβληματισμοί παρά οτιδήποτε σίγουρο. Η πρόοδος λοιπόν, πώς βλέπουμε την πρόοδο, πώς μπορούμε να συνεχίσουμε. Μπορώ να συνοψίσω λέγοντας ότι η πρόοδος ε, είναι αρκετά καλή. Υπάρχει ένα θέμα ετοιμότητας πριν από οποιαδήποτε επιχείρηση, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και οι διάφορες πρωτοβουλίες που λαμβάνουν χώρα μέσω διαρθρωμένου διαλόγου πάνε καλά. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να σημειωθεί πρόοδος ιδιαίτερα τέτοια, σε τέτοια εποχή κρίσης και βλέπω ότι η ζωή ε, συνεχίζεται παρά τις ε, διάφορες αναβολές ε, λοιπόν. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι υπέρ της πρωτοβουλίας E2I των 8 ομάδων εργασίας χωρισμένων σε γεωγραφικές ζώνες. Νομίζω ότι η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι οι μόνε χώρε που συμμετέχουν σε κάθε μία από αυτέ τι ομάδε εργασία. Δείχνει λοιπόν αυτό πόσο σοβαρά παίρνουμε το θέμα αυτό. Επίσης συμμετέχουμε σε άλλους ε, οργανισμούς ε, και στον ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπουδήποτε υπάρχουν ε, θέματα ασφάλειας προς Η συμμετοχή μας λοιπόν στα διεθνή φόρα έχει τύχει πλήρου στήριξη από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η πρόοδος που έχει σημειωθεί είναι αρκετά καλή. Ενώ σας άκουγα, έχω σημειώσει κάποια θέματα τα οποία με βρίσκουν σύμφωνο, δηλαδή συμπληρωματικότητα, συνέργεια, διαφάνεια, όλα αυτά είναι και για μας πάρα πολύ σημαντικά, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι επιδόσεις μας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει καλή επικοινωνία έτσι ώστε να υπάρξει μια καλή συνεργασία. Τώρα υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες που καλύπτουν το θέμα της ετοιμότητας μέσω διάφορων ε, ομάδων, μέσω ε, διαφόρων ε, βημάτων που ασχολούνται με θέματα ετοιμότητας, με διάφορες ασκήσεις οι οποίες ε, έχουν θέμα αποτρεπτικό και είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει καλή συνεργασία και καλή επικοινωνία έτσι ώστε να αξιοποιηθούν στο έπακρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ βασικός παράγοντας λοιπόν που δένει τις προσπάθειες όλων αυτών των κρατών μελών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις συνέργειες μεταξύ πρωτοβουλειών η E2I μία από αυτές τις πρωτοβουλίες. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε πόσο σημαντική είναι η συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Είναι σημαντικό επίσης τα φόρα να μην είναι υπέρ το δέον έτοιμα να περιγράψουν τις ε, αρμοδιότητες του καθενός. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να εθετήσουμε μία προσέγγιση βασισμένη σε αρχές μια ρεαλιστική προσέγγιση που θα πρέπει να είναι στόχος του στρατιωτικού προσωπικού κατά την προετοιμασία των ε, ενόπλων δυνάμεων. Και νομίζω πως έχουμε συζητήσει στο παρελθόν ε, πάλι το αν η συγκέντρωση δυνάμεων είναι ε, μια καλή ιδέα και πώς και πού θα έπρεπε να γίνει αυτό. Το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρεί πως ε, αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Το E2I, και θα το τονίσω αυτό, ε, δεν έχει στρατιωτικό χαρακτήρα. Είναι μια συνάντηση που λαμβάνει η χώρα σε ένα κλειστό χώρο, υπάρχει ανταλλαγή απόψεων, δεν υπάρχει κάποια κοινή στρατιωτική επιχείρηση. Μας περιορίζει λοιπόν η εντολή μας και προτού γίνει οποιαδήποτε επιχείρηση στο έδαφος χρειάζεται επικοινωνία και οργάνωση έτσι ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε όπως θα έπρεπε. Η E2I λοιπόν είναι μια ε, τέτοια δυνατότητα αποτελεί ένα τέτοιο ε, φόρουμ. Τώρα, νομίζω πως ε, δεν υπάρχει κάποια ανησυχία να περάσουν ορισμένα, ορισμένες επιχειρήσεις την εντολή τους. Χρειάζεται να εξετάσουμε διάφορα σενάρια και να δούμε όλες τις ε, δυνατότητες που έχουμε. Υπάρχει το κέντρο ανάπτυξης ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, κέντρο ανάπτυξης ε, δόγματος. Υπάρχει και ένα αντίστοιχο κέντρο στη Γερμανία. Προσπαθούμε λοιπόν να ανταλλάσσουμε πληροφορίες και να συνεργαστούμε προτού δημοσιοποιήσουμε οτιδήποτε. Το DCDC στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως είπε και ο Γάλλος συνάδελφος, ε, έχει εκπροσώπους από ε, πολλές χώρες, από τη Γαλλία, από τη Φιλανδία. Υπάρχει το MCDC, η ομάδα που στηρίζεται και από τις Ηνωμένε Πολιτείε, ασχολείται με θέματα ανάπτυξης και νομίζω πως ε, υπάρχουν πολλά φόρα που ήδη εξετάζουν διάφορα σενάρια, ήδη εξετάζουν τις βέλτιστες πρακτικές και δεν ξεκινάμε λοιπόν από το τίποτα. Έχουμε υλικό πάνω στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε. Νομίζω πως η E2I θα χτίσει πάνω σε αυτό το υλικό και θα έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε και στο μέλλον, μέσω του ΝΑΤΟ ή μέσω κάποιου άλλου φόρουμ. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Δίνω το λόγο τώρα στο στρατηγό. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λέγομαι Wolfgang King. Είμαι εκπρόσωπος στρατιωτικός ε, της Στρατιωτικής Επιτροπής ε, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε σε αυτούς τους χώρους εκπροσωπώ τις γερμανικές θέσεις. Υποστηρίζουμε την πρωτοβουλία αυτή που παρουσίασε ο Γαλλός ε, συνάδελφος και χαίρομαι που μπορώ να είμαι εδώ σήμερα ε, με τους, ε, αυτούς που επινόησαν αυτή την πρωτοβουλία από γερμανικής πλευράς. Εμείς συνεργαζόμαστε και έχουμε δεσμευτεί για αυτή την πρωτοβουλία διότι θεωρούμε ότι ό,τι έχει να κάνει η Ευρώπη στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής ε, και πολιτικής ασφάλειας ε, εξυπηρετεί και τα γερμανικά συμφέροντα. Αυτή η πρωτοβουλία είναι το κατάλληλο φόρουμ, κατά την άποψή μας, ούτως ώστε ε, εν τέλει να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών, συντονισμό και δικτύωση. Όπως είπε μόλις ο Βρετανός συνάδελφος. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε και στι δύο πρωτοβουλίε που ανέφερε ο Γάλλος συνάδελφο θα πρέπει να έχουμε λιγότερες επιχειρησιακές ε, ε, διαστάσεις, αλλά να δούμε περισσότερο πώς θα προωθήσουμε τα δομικά κομμάτια. Δεν έχουμε αντίθετη θέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Αντιθέτως, ε, κοιτάμε να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τα πράγματα και να βελτιώσουμε τα πράγματα και να επιτυχούμε περισσότερα. Το ζήτημα της προόδου είναι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μας. Η πρωτοβουλία αυτή δεν πρέπει να δημιουργήσει κάποιο αποκλειστικό χώρο θα θέλαμε να συμμετέχουν και άλλα κράτη και θέλουμε να υπάρχει διεύρυνση και χαιρόμαστε που υπήρξε διεύρυνση ήδη ώστε να, έχουμε, να ακολουθούμε συγκεκριμένες διαδικασίες με τα νέα μέλη και να ακολουθούμε ε, συγκεκριμένες διαδικασίες. Χωρίς να αναλύσω την πρωτοβουλία, γιατί σίγουρα θα έχετε πολλές ερωτήσεις, θα πω εν συντομία, εμάς μας ενδιαφέρει να ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση μας ενδιαφέρει στον τομέα αυτόν να ενισχύσουμε την πολιτική ασφαλεία τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Όλα όσα σχετίζονται με αυτά ε, εξυπηρετούν τα συμφέροντά μας. Ε, η υποστήριξη αυτή λοιπόν δεν αποτελεί ε, αντίθετη θέση από γερμανική πλευρά έχω να πω ότι όσον αφορά την άμυνα τη Ευρώπη κατά κάποιο επιτιθέμενο εξωτερικό θα το πει καθαρά και ο Εστονός συναδελφός, ε, η Ευρώπη θα πρέπει να είναι ο σύμμαχος που είναι αυτή τη στιγμή το ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ. Merci, euh, le Merci. Σας ευχαριστώ και ο συνταγματάρχης Ρίκαρντ. Καλημέρα σε όλους. Είμαι ο συνταγματάρχης Ρίκαρντ. Ε, Είμαι τετραμένος στη Γαλλία, στην Ισπανία και ασχολούμαι με επιχειρησιακά θέματα και θέματα EI2. Πολλά υπόθηκαν ήδη για την EI2. Δεν θέλω να επαναλάβω πράγματα που υπόθηκαν για την Εστονία. Σίγουρα η EI2 είναι ένα σημαντικό πλαίσιο συνεργασίας που συγκεντρώνει τα κράτη-μέλη της Ευρώπης που επιθυμούν να ανταποκριθούν μαζί σε απειλές και σε κρίσεις για την ασφάλεια των πολιτών μας. Η στενή συνεργασία και ο συντονισμός ε, για δραστηριότητες τέτοιες είναι σίγουρα σημαντικό. Είναι πιο αποτελεσματική ανταπόκρισή μας ε, αν ανταποκρινόμαστε κοινά σε κοινέ απειλέ. Κατά τη δική μας άποψη λοιπόν πρόκειται για ένα φόρουμ πολύ καλό ε, όπου μπορούμε ανοιχτά να συζητήσουμε και ελεύθερα όλα τα ζητήματα. Δεν υπάρχουν πολιτικά όρια σε αυτό τον κλάδο. Η ασφαλή της Εστονίας είναι ασφάλεια και της Ευρώπης ε, και είναι σημαντικό να το αναφέρουμε. Και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ η Εστονία συμμετείχε σε δύο ομάδες εργασίας Είμαστε μέλος της ασφάλειας στη Βαλτική και στην, ε, συμμετέχουμε και στην ομάδα εργασία για το ΣΑΧΕΛ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Ήδη πέρυσι ξεκινήσαμε ε, διμερείς ε, στρατιωτικές επιχειρήσεις με τη Γαλλία στο ΣΑΧΕΛ και το φόρουμ αυτό αποτελεί μια εξαιρετική πλατφόρμα ε, ανταλλαγής πληροφοριών. Επειδή εγώ ασχολούμαι με αυτά τα ζητήματα ΙΑΕΤΟΥ σε πρακτικό επίπεδο, και όχι πολιτικό. Έχω να πω ότι βλέπουμε πολύ καλό μέλλον για το φόρουμ αυτό. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να ξέρω αν κάποιο από τα μέλη θα ήθελε να παρέμβει στη συζήτηση, αν θα ήθελε να έχει το λόγο. Monsieur Peters. Ο κύριος Peters. Oui, Madame Chair, uh, dear Πρόεδρε, Σταδηγή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Είναι προφανές ότι η πρωτοβουλία της Γαλλίας είναι πάρα πολύ σημαντική έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Άμυνα να καταστεί βαρότερη. Όπως είπατε, πολλές χώρες έχουν συμμετάσχει στην πρωτοβουλία αυτή, η οποία είναι καλή. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχει και η ΠΕΣΚΟ. Μία πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε βάσει του άρθρου 24, παράγραφος 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο γνωρίζετε φυσικά. Ποια όμως είναι η σχέση μεταξύ ΠΕΣΚΟ και της πρωτοβουλίας που μας αναφέρατε. Υπάρχουν κάποιες ε, ερωτήσεις που προκύπτουν. Υπάρχουν κάποια μέλη που, ε, δεν, που είναι ε, μέλη στην μία πρωτοβουλία και όχι στην άλλη. Η Δανία, για παράδειγμα. Και αυτό μου φαίνεται κάπως παράξενο. Έπειτα, νομίζω πως Ίσως θα ήταν καλύτερο να γίνει μια συγχώνευση των ε, δύο πρωτοβουλειών, διότι χρειάζεται να έχουμε ευρωπαϊκή άμυνα και μια πολιτική πιο ισχυρή από ό,τι στο παρελθόν. Όμως η ύπαρξη ταυτόχρονα δύο διαφορετικών πρωτοβουλειών θεωρώ ότι αποδυναμώνει κάπως την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπειτα αναφερθήκατε στο ΝΑΤΟ και γνωρίζω βέβαια ότι η πρωτοβουλία αυτή αποδυναμώνει μεν το ρόλο του ΝΑΤΟ, όμως θα δώσει και ένα ισχυρό μήνυμα ότι τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία ψάχνουν ένα μήνυμα. Ποιο είναι λοιπόν το μήνυμα που στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο ΝΑΤΟ με αυτό. Σας ευχαριστώ. Ας ακούσουμε κάποιες ερωτήσεις πρώτα και μετά θα απαντήσετε από εκείνο. Ο κύριος Στρεβίσιους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Ε, είναι η πρώτη φορά που μιλούμε για την ε, πρωτοβουλία αυτή παρέμβασης και επομένως ε, ακούγεται πολύ ενδιαφέρον και πολύ καινούριο. Ακούω τις λέξεις συμπληρωματικότητα και συνέργεια ποιος είναι ο συσχετισμός με την ε, ομάδα, την, το battle group της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέλος πάντων. Ε, θα υπάρξει κάποια συμπληρωματικότητα προς τη μονάδα αυτή. Γιατί περιμέναμε να δούμε κάποια νεότερα σχετικά με αυτό. Τώρα, επίσης, σε περίπτωση ε, Brexit, οι χώρες εταιρικής σχέσης θα μπορούν να έχουν πλήρη συνεργασία και συμμετοχή σε αυτήν την κοινή στρατιωτική δύναμη στο μέλλον. Γιατί και άλλες χώρες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συνεργασίας. Γιατί η εταιρική σχέση βεβαίως είναι κάτι πολύτιμο, ιδιαίτερα στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας και της πρωτοβουλίας. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο στους αξιωματικού που επιθυμούν να απαντήσουν σχετικά με τα ερωτήματα που επιθυμούν να απαντήσουν όπως θέλετε εσείς. Ευχαριστώ Πρόεδρε για πολύ ενδιαφέρουσες ε, ερωτήσεις με συγχωρείτε, για την ε, ΠΕΣΚΟ, την μόνιμη αυτή δομή. Η δια, διεπιχειρησικότητα, διαλειτουργικότητα προκύπτει από τις δοκιμές ε, αλλά και την ανταλλαγή πρακτικών, γνώσεων, δεδομένων κτλ. Ε, έτσι αναπτύσσεται ένα αμυντικό ή ένα στρατιωτικό δόγμα και οι συζητήσει στις τέσσερις βασικές θεματικές ε, ε, μας βοηθάει να καταλάβουμε τι μπορεί ο καθένα να κάνει καλύτερα και πώς μπορούμε να συνεργαστούμε. Η διαλειτουργικότητα ε, προποθέτει να έχουμε τις λιγότερες δυνατές, τα λιγότερα δυνατά εμπόδια όταν επιθυμούμε να αναλάβουμε δράση. Επομένως, αν μια ομάδα ή μια οργάνωση ή μια δομή είναι υπερβολικά εξαντλητική στους κανόνες της, αυτό επιβάλλει όρια στην διαλειτουργικότητα που προσπαθούμε να επιτύχουμε. Περιορισμό των δυνατοτήτων, του εξοπλισμού μας, των κοινών μας ε, ε δοκιμών και ασκήσεων. Επομένως, εάν η μόνιμη δομή ασφαλείας επιθυμεί να παράσχει ένα πλαίσιο καθότι λειτουργούμε στον αμυντικό τομέα όπου ο ρεαλισμός είναι ίσως πιο σημαντικός από τις αρχές και τις αξίες λέει ο Μιλτής όταν έχουμε μια πραγματική δουλειά να κάνουμε και επομένως όσο λιγότερο αυστηροί είμαστε σε ένα πλαίσιο κανονιστικό τόσο καλύτερες δυνατότητες προσφέρουμε στις ε, χώρες που συμμετέχουν. Για την στρατιωτική δύναμη, ε, για το battle group που αναφερθήκατε, ε, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει συμμετάσχει με παροχή δυνάμεων. Σήμερα έχουμε δυνάμεις από χώρες που δεν είναι καν κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορούν να συνεισφέρουν δυνάμεις σε αυτή τη δέσμη επιχειρησιακή ετοιμότητα του Battle Group και επομένως υπάρχει προηγούμενο και υπάρχει και η δυνατότητα στο μέλλον κράτη μη μέλη να μπορούν να συμμετάσχουν. Ελπίζω να έχω απαντήσει στην ερώτησή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συμπληρωματικά ως προς τα όσα είπε ο Βρετανός συνάδελφος για την πρώτη ερώτηση, εξαιρετική κυρία. Απαντήσατε εσείς ο ίδιος όταν είπατε ότι η Δανία πράγματι ε, έκανε opt-out ε, από την ΠΕΣΚΟ, το Ηνωμένο Βασίλειο με το Brexit. Ε. δεν θα συμμετέχουν σε αυτήν την πρωτοβουλία, θα ήταν περίπλοκη η συμμετοχή τους, οπότε τουλάχιστον αυτό έχει λήξει. Σίγουρα δεν είμαστε στην ΠΕΣΚΟ για να θέλουμε μόνο μέλη των Ευρωπαϊκή ε, της Ευρωπαϊκής Ένωση, οπότε ε, θεωρούμε ότι η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασίλειου και τη Δανία ήταν σημαντική. Θέλουμε τι σημαντικέ χώρε. Ο δεύτερο λόγο είναι πιο σημαντικό ακόμα. Τα εργαλεία αυτά δεν κάνουν το ίδιο πράγμα. Πίσω από αυτές τις δύο πολιτικές υπάρχει στρατηγική κοινή, η στρατηγική αυτονομία, αυτή η έννοια. Είναι δύο μέσα όμως πολύ διαφορετικά. Ε, στο πλαίσιο μιας ε, περιορισμένης ομάδας που έχει ήδη ένα σημαντικό κοινό ε, χαρακτήρα το στρατηγικό, γι' αυτό επέλεγε να γίνει και όπως υπενθύμισε ο Βρετανός συνάδελφος χωρίς την αυστηρότητα που απαιτεί η συνένεση στα ευρωπαϊκά όργανα για παράδειγμα έτσι θεωρούμε ότι θα είναι πιο εύκολο να επιτυγχάνουμε και να αναπτυσσόμαστε προς όφελος Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και προς όφελος του ΝΑΤΟ αυτή την κοινή στρατηγική. Και το ωφέλη της αυτό θα επηρεάσει, θεωρούμε θετικά, και τους θεσμούς και εκτός. Αυτή η κοινή ε, στρατηγική κουλτούρα ε, οικοδομείται μέσω αυτού του επιχειρησιακού πνεύματος. Αυτό που ονομάζουμε horizon scanning, δηλαδή προσπαθούμε να καταλάβουμε πού ζούμε σε ένα φόρουμ αρκετά περιορισμένο. Μπορούμε να κάνουμε και τι ανταλλαγέ σε πολύ καλά ε, σε ένα πολύ καλό επίπεδο, απόρριτο χωρίς ε, ψημαχίες συναισθηματικές, ε, μπορούμε να ασχοληθούμε με ζητήματα που δεν θα μπορούσαν οι χώρες αρχικά να, να προγραμματίσουν και τέλος δημιουργούμε δεσμούς, επαφές, εμπιστοσύνη. Πάντα, όπως είπα, είναι ευκολότερο σε, στο πλαίσιο τόσο μικρών ομάδων. Τώρα για το EU Battle Group. Μην ξεχνάτε, ειλικρινά το λέω και υπενθυμίζω αυτό που βρεταν ο συνάδελφος προηγουμένως, ότι πρόκειται για ένα φόρουμ. Δεν είναι δύναμη το ei Και ελπίζω ότι θα έχει ως αποτέλεσμα κάποια στιγμή να αξιοποιείται καλύτερα η ευρωπαϊκή μάχη με δύναμη, διότι θα υπάρχει μια κοινή στρατηγική κουλτούρα, η οποία θα έχει φτάσει σε κάποια τελική μορφή από αυτές τις 10 χώρες, ε, η οποία θα διαπνεύσει τελικά την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ε, μπορέσουμε έτσι να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα αυτό το EU Battle Group. Ευχαριστούμε. Ε, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Νομίζω πως ε, αναφερθήκατε ακριβώς σε αυτά που απασχολούν και τους ε, Γερμανούς βουλευτές, δηλαδή γιατί ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Ε, δεν θέλουμε να αντικαταστήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο ΝΑΤΟ, αυτό σας το υπογράφω. Η ομάδα μας συναντιέται μία φορά την εβδομάδα, ανταλλάσσει απόψεις, προετοιμάζει τις επόμενες συνεδριάσεις, όμως ο κύριος ε, στρατηγικός σχεδιασμός λαμβάνει χώρα στα Υπουργεία. Και αυτό αποτελεί ε, προστιθέμενη αξία από μόνο του. Τα θέματα αυτά τα οποία μας απασχολούν και απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, εμένα και εσάς, είναι θέματα τα οποία απασχολούν και αυτό το δίκτυο. Και είναι πλεονέκτημα να υπάρχει ένα δίκτυο συνεργασία έτσι ώστε να μπορούμε να ανταλλάσσουμε απόψεις ε, και δεν έρχεται σε καμία περίπτωση σε αντίθεση με τις επιτροπέ αυτές. Το γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι η σύσταση μια τέτοια ομάδας δεν είναι στρατιωτική ε, ενέργεια, είναι κάτι που δηλώνει την πολιτική βούληση, δηλώνει πώ έχουμε ε, κάποιου κοινού στόχου. Τώρα, η διατύπωση intervention, δηλαδή παρέμβαση, είναι μια διατύπωση η οποία έχει τονιστεί στον γερμανικό τύπο, έχει αναφερθεί ότι έχει μεγάλη βαρύτητα, βέβαια. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι παρουσιάζει ο τύπος σε ό,τι αφορά την ε, πρωτοβουλία αυτή. Και ξέχασα να πω κάτι άλλο που με ενδιαφέρει προσωπικά. Στη Μαύρη Θάλασσα υπάρχει μια περιοχή που ε, δεν συμπεριλαμβάνεται στο πεδίο δράσης. Είναι μια περιοχή την οποία χειρίζεται το ΝΑΤΟ Επιχειρούμε λοιπόν εμείς, όπως σας είπα από την αρχή, να επιλέξουμε ομάδες εργασίες που να μην έχουν επικάλυψη με άλλες εργασίες ή άλλες συνεργασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, επομένως, η Μαύρη Θάλασσα είναι ένα θέμα νατοϊκό, αν θέλετε να το πούμε έτσι. Ευχαριστώ όλους. Αν δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη του πάνελ για τη διαθεσιμότητά τους σήμερα.

Euh, λοιπόν, επειδή λείπουν τα περισσότερα μέλη της υποεπιτροπής,